Καλώς ορίσατε αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε παρακαλώ. και κύριοι, κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Γεωργίας. Ε, με βασικό θέμα της πρωινής ημερήσιας διάταξης την Σλοβακική Προεδρία. Έχουμε την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, την Υπουργό Γεωργίας της Σλοβακίας. Θα κάνω ιδιαίτερα το χαιρετισμό της αργότερα. Ας δούμε πρώτα όμως κάποια διαδικαστικά. Ως προς την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω της απουσίας της κυρίας Γκέρλινγκ, το 10, δηλαδή ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών, την οδηγία ΝΕΚ δηλαδή, το σημείο αυτό αναβάλλεται για τις 26 Σεπτεμβρίου. 26 Σεπτεμβρίου, το σημείο 10 της κυρίας Γκέρλινγκ. Με αυτή την αλλαγή μπορούμε να κρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ωραία. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Σημείο 2. Να σας πληροφορήσω ότι τον κύριο Βοητσεχόφσκι που ανέλαβε πολύ σημαντικά καθήκοντα σε άλλο κοινοτικό θεσμικό όργανο αντικαθιστά η κυρία Ούρσουλα Κρούπα την οποία και καλωσορίζουμε θερμότατα. Η κυρία Ούρσουλα Κρούπα ε, ήδη ήταν Ευρωβουλευτής στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία 2004-2009 Καλώς ήρθατε και πάλι κυρία Κρούπα. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ανάληψη των καθηκόντων σας. Ήδη έχετε πλούσια εμπειρία και ε, υπολογίζουμε και στη δική σας συμμετοχή και συνεισφορά στην Επιτροπή μας. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 21 γλώσσες με εξαίρεση τα εσθονικά, μαλτέζικα και γοεδελικά. Και επίσης ε, η συνεδρίασή μας αναμεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Θα ήθελα τώρα να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 24ης Μαΐου και 6ης Ιουνίου 2016 με τη συνήθη διαδικασία. Όπως σας είπα, το κυρίως θέμα της πρωινής μας συνεδρίασης είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Προεδρία του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου Γεωργίας, την Υπουργό Γεωργίας της Σλοβακίας, την κυρία Γκαμπριέλα Ματετσνά. Είχαμε και συνάντηση εργασίας ήδη σε επίπεδο συντονιστών, οπότε γνωρίζουμε την κυρία Υπουργό. Σας καλωσορίζω θερμότατα και σας ε, ενημερώνω ότι περιμένουμε ιδιαίτερος ε, και με πολύ ενδιαφέρον την ανταλλαγή απόψεων και την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Σλοβακικής Προεδρίας. Και περιμένουμε τις απόψεις για πολλά σημαντικά θέματα που λαμβάνουν χώρα. Για παράδειγμα το μέλλον της κοινής γεωρικής πολιτικής, η απλούστευσή της, τριμερείς διάλογοι για τη βιολογική γεωργία, πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις, επίσης την κρίση σε πολλές γεωργικές αγορές. Το γνωρίζετε κύριε Υπουργέ. Και μάλιστα τη Δευτέρα προεδρεύσατε στο Συμβούλιο Γεωργίας και εκεί ακούσατε τον Επίτροπο Χόγκαν που μίλησε για τις δράσεις που θα αναλάβει στο γαλακτοκομικό τομέα. Και ε, στις 19 Ιουλίου θα έχουμε και την σχετική ενημέρωση. Ε, όσοι ήθιστε, αμέσως μετά τη δική σας ομιλία θα λάβουν το λόγο συντονιστές. Και μετά από αυτή την αρκετά μακροσκελή εισαγωγή ήρθε η ώρα να σας δώσω το λόγο. Σας καλωσορίζω και πάλι εγκαρδιότητα, εγκαρδιότητα και σας δίνω το λόγο κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια με τα οποία με καλωσορίσατε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσοι δέχτηκαν την πρόσκλησή μας ε, στο σύντομο πρωινό εργασίας που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο και για τις δύο πλευρές. Όλοι μπορέσαμε να ακούσουμε τα βασικά μας θέματα και τις προτεραιότητες ε, όπως τα παρουσιάσαμε και με ενδιαφέρον άκουσα και τις απόψεις των έρετων ε, μελών αυτού του Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου λοιπόν κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτές να σας πω δύο λόγια σήμερα. Η Σλοβακική Δημοκρατία αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον τομέα της Γεωργίας επίσης και θεωρούμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως σημαντική συνιστόσα της εργασίας μας. Θέλουμε να επιδιώξουμε να βρούμε λύσεις σε προβλήματα μαζί σας και να ε, δώσουμε αποτελέσματα υποφιλή για τους πολίτες, τους ε, αγρότες, ε, τις επιχειρήσεις ε, σε ολόκληρη την Ένωση. Η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την ελκυστικότητα του τομέα της γεωργίας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια αλλαγή γενναιών. η παρούσα Επιτροπή είναι βασικός εταίρος και θα μας βοηθήσει να τα πετύχουμε όλα αυτά. Η Σλοβακία αναλαμβάνει την Προεδρία σε δύσκολες εποχές. Μόλις είχαμε το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι γεωργοί έχουν να αντιμετωπίσουν την αστάθεια στις αγορές, έχουμε την κλιματική αλλαγή και την ε, οικονομική κρίση που συνεχίζεται, το ρωσικό εμπάργκο. και ο γαλακτοκομικό τομέα, ε, οι μεγάλοι γεωργικοί τομεί ε, οι τομείς των φρούτων και των λαχανικών δεν σημειώνουν πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη, παρότι στο γαλακτοκομικό τομέα με την έλευση τη κρίση. Ε, παρότι αναμένονταν πολλά προβλήματα, η κρίση αυτή διήρξε περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Ωστόσο, καταφέραμε να μετριάσουμε τι επιπτώσει αυτή τη κρίση. Αλλά μάθαμε ένα πράγμα το γάλα είναι ένα πολύ ευαίσθητο αγαθό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσει τους πρωτογενείς παραγωγούς τροφίμων. Ε, αν μη τι άλλο, διότι αποτελούν βασική συνιστόσα στις αγροτικές περιοχές. Βλέπουμε πως η γεωργία αντιδρά σε εξωτερικά ερεθίσματα και η αυξημένη προστασία του τομέα αυτού είναι κάτι αναγκαίο. Εμείς ως Προεδρία θα παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στις αγορές, στις αγορές γεωργικών προϊόντων. Και ευχαρίστω ε, να συζητήσουμε οποιοδήποτε ζήτημα στο Συμβούλιο Υπουργών. Το Συμβούλιο θα αξιολογεί τις ε, πληροφορίες που λαμβάνει. Εδώ και καιρό λέμε ότι χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή λύση στον τομέα αυτών, βασισμένη στην αρχή της αλληλεγγύης. Τι έδειξε η σημερινή κρίση, ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία της ε, τροφικής αλυσίδας. Μακροπρόθεσμη προτεραιότητα της Σλοβακίας είναι η καθιέρωση δίκαιων σχέσεων στην τροφική αλυσίδα. Θέλουμε να αυξήσουμε τη διαφάνεια του συστήματος και να παρεμποδίσουμε ε, πρακτικές, αθέμητες πρακτικές ανταγωνισμού. Έτσι η Σλοβακία θέλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της βελτίωσης ε, της θέσης των αγροτών στην τροφική αλυσίδα. Καλωσορίζω λοιπόν την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της έκθεσής του που εγκρίθηκε τον Ιούνιο φέτος. να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις εξαιρετικές προσπάθειες που έγιναν ε, για να λάβει αυτή η εκθέση την τελική της μορφή. Η συνεργασία με τρίτες χώρες σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο είναι κάτι σημαντικό. Ωστόσο, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της αποδέσμευσης των αγορών και της προστασίας των αξιών της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των διεθνών διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δημιουργήσουμε χώρο για την προετοιμασία των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών όπως TTIP, Mercosur ή οποιονδήποτε άλλων μελλοντικών συμφωνιών με τρίτες χώρες που ενδέχεται να προκύψουν. Η επικύρωση των συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών ωστόσο πρέπει να θεωρείται στο πλαίσιο κρίσιμων συνθήκων ε, στις ευρωπαϊκές αγορές γιατί οι ευρωπαϊκές αγορές ε, δυσκολεύονται να απορροφήσουν ε, όλες τις ποσότητες βασικών αγαθών. Οπότε αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ όταν πρόκειται να υπογράψουμε συμφωνίες τέτοιες με τους εταίρους μας. Τώρα για το θέμα της απλούστευσης της κοινή γεωργικής πολιτικής θα ήθελα να εστιαστώ στα ζητήματα εκείνα όπου υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα μείωση της γραφειοκρατίας τόσο για τους αγρότες όσο και για τις αρχές. Είμαστε επεπισμένοι ότι η ύπαρξη της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής ε, αιτιολογείται επαρκώς. Μπορεί να αποτελέσει μια καλή απάντηση για τις προκλήσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Όχι μόνο όσον αφορά την αηφορία της παραγωγής, την ε, διατροφική ασφάλεια, αλλά και διότι θα βοηθήσει να διατηρήσουμε το ε, χαρακτήρα της, ε, της Ευρωπαϊκής Γεωργίας ε, και των περιοχών της Υπέθρου. Η Σλοβακική Προεδρία θα συνεχίσει το έργο της Ολλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό για τη βιολογική γεωργία και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Στόχος αυτού του κανονισμού είναι να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στους ε, βιολογικούς γεωργούς και η απλούστευση της μετάβασης ε, στη βιολογική παραγωγή για όλο και περισσότερους αγρότες. Εμείς πιστεύουμε ότι η βιολογική γεωργία θα αποτελέσει την εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής ε, Γεωργίας. Χρειάζεται ένα καλά δομημένο και σταθερό πλαίσιο ώστε να αναπτυχθεί και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά της. Ένα άλλο σημείο που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι η δασοκομεία. Θα το αναφέρω και αργότερα στην ομιλία μου, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η δασοκομεία και τα δάση μπορούν να επηρεάσουν ε, σημαντικά θετικά μάλιστα τις λύσεις που θα δοθούν για την αντιμετώπιση των σημερινών κλιματικών αλλαγών, των προβλήματων βιοποικιλότητας και αηφόρων ανάπτυξη γενικότερα. Λόγω αυτού είναι αυξημένε οι απαιτήσει ε, προς τα ευρωπαϊκά δάση, οι οποίες μεταφράζονται σε διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες, σε διάφορους τομείς. Τι θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλουμε η δασοκομεία να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά σημεία στο Συμβούλιο, των συζητήσεων στο Συμβούλιο ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να αξιοποιηθεί ο πολυλειτουργικός ρόλος των δασών και να καθοριστεί ένα διεθνές πλαίσιο για την αηφόρο διαχείριση των δασών. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σε ε, διεθνείς ε, πολυμερείς οργανισμούς όπως ε, ο Διεθνής Οργανισμός, οι Διεθνείς Οργανισμοί για τα Δάση σκοπός μας είναι να επιτύχουμε μια κοινή, να επιτυχάνουμε κοινέ θέσει που θα ανταποκρίνονται σαφώ στι απόψει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών όσον αφορά τι σημερινέ εξελίξει ε, στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαλόγου για τα δάση και τη δασοκομεία. Τώρα όσον αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα και την ε, διατροφική ασφάλεια, στι δραστηριότητε μα έχουμε διασφαλίσει και θα συνεχίσουμε να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε νομοθεσία εκπονείται, εφαρμόζεται ολοκληρωμένα. Εδώ έχουμε μία δέσμη μέτρων πολύ σημαντική, περιλαμβάνει δύο προτάσεις. Μία πρόταση για τις φαρμακούχες ζωοτροφές και μία για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Όσον αφορά τις φαρμακούχες ζωοτροφές, στην πρόταση αυτή θέλουμε να ολοκληρωθούν οι τεχνικές συζητήσεις για το έγγραφο αυτό στο Συμβούλιο και πρέπει να πω ότι έχουν προχωρήσει αρκετά οι συζητήσεις εδώ. Έχουμε αντίληψη και ε, συνέστη του σκοπού για τον οποίο έχει εκπονηθεί αυτό το νομοθέτημα. Ένας από τους πολύ σημαντικούς και ενδιαφέροντες τομείς για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η χορηγήση φαρμακούχων ζωοτροφών σε ζώα. Αλλά πρέπει να πω ότι η οριστικοποίηση αυτού του θέματος θα βασιστεί στην ολοκλήρωση της πρότασης ε, για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Είναι σε αυτές οι δύο προτάσεις. Παρότι η Κομάγκρη δεν είναι η βασική επιτροπή, η επιτροπή, επιτροπή για αυτά τα δύο θέματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι γνωμοδοτήσει τη επιτροπής αυτής ε, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων που θα λάβει χώρα το Μάρτιο. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί δηλαδή το θέμα αυτό, αλλά θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, ενδελεχείς και να συμμεθεί πρόοδος ε, στις συζητήσεις επί αυτών των προτάσεων στο Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω κυρίε και κύριοι ότι έχουμε την πρόθεση να καταπολεμήσουμε την μικροβιακή αντίσταση. Πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία, αλλά θέλουμε να μεριμνήσουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει υψηλά πρότυπα για την προστασία τόσο της υγείας των ζώων όσο και της υγείας των ανθρώπων. Όσον αφορά τον κανονισμό περί επισήμων ελέγχων, όπου έχει, για τον οποίο έχει εκπονήσει γνωμοδότηση επίσης η Κομάγκρη, έγινε μια ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή της Ουσίας στην ΕΜΒΗ χθες, η οποία ενέκρινε την γνωμοδότηση αυτή. αφού ψηφίσει και στην Ολομέλεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θελήσουμε να διασφαλίσουμε την υλοποίηση αυτή στις νέες νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τομεί ε, όπου θέλουμε να παρακολουθούμε την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τι μολύσει, την κτηνοτροφία, την καλή μεταχείριση των ζώων, τη συνεργασία με τρίτε χώρε, τις ε, συνθήκες ε, εξαγωγών και εισαγωγών αλλά και την πρόσβαση στις αγορές και θα θέλαμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για την πρόληψη της απάτης των τομέα των τροφίμων και θα θέλαμε να αναθεωρήσουμε και την έκθεση της Κομισιόν που σχετίζεται με μια γενική διατροφική νομοθεσία και το ζήτημα της επαλήθευσης του συστήματος ελέγχου που έχει προβλεφθεί από την Κομισιόν και που στοχεύει στο να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την επιβολή τη και την εφαρμογή τη. Ένα άλλο τομέα στον οποίο θέλουμε να εστιαστούμε είναι το σχέδιο κανονισμού για τα λοιπάσματα. Αυτό θα πρέπει να ανοίξει την αγορά για καινοτομίε. Αποτελεί κομμάτι μια δέσμη μέτρων που αφορά την ανακύκλωση. Εμεί θέλουμε να συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει και να μελετήσουμε τι δυνατότητε ανάπτυξη μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο. Τέλος, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο υπό τη Σλοβακική Προεδρία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων αγροτών. Θα επιδιώξουμε να βρούμε λύσεις που θα συμβάλλουν στη σταθερότητα του τομέα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι και εγώ η ίδια θα προσπαθήσω να πω σε όλους μας τους πολίτες ότι η γεωργία είναι ένας τομέας που συμβάλλει σημαντικά στην υγεία όλων μας. Είναι όμως επίσης και ένας τομέας που παρέχει πολλές θέσεις εργασίας σε πολλοί κόσμο και ειδικότερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης ένας τομέας ε, που μπορεί να απορροφήσει ε, πολλές νέες καινοτομίες. Θα, θα πω στους Ευρωπαίους ότι η γεωργία είναι ένας τομέας ο οποίος επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να συμβάλλει και στο μετριασμό της κλιματικής αναλλαγής και μπορεί να συμβάλλει και στην ανάπτυξη που είναι τόσο απαραίτητη για όλες τις χώρες μας. Η γεωργία και οι εργαζόμενοι στον τομέα της γεωργίας αξίζουν την εμπιστοσύνη μας, το ενδιαφέρον μας και τη βοήθειά μας. Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω όλους ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε λύσεις σταθεροποίησης του τομέα. Και τέλος, θα ήθελα να παραθέσω την κυρία Μάρλεν Τίμερμαν, Ολλανδή γιατρός και πολιτικός, που λέει ότι σε αυτές τις προσπάθειες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καλός πολιτικός είναι αυτός που συνδέει τους ανθρώπους για την ευημερία των λαών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Πολύ εκτενής ε, και περιεκτική η παρουσίαση των προτεραιοτήτων και των πρωτοβουλειών της ε, Σλοβακικής Προεδρίας. Και όπως ε, σας είπα και προηγουμένως, θα ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές και μετά του, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Δύο λεπτά θα έχει ο κάθε συντονιστής στη διάθεσή του και ένα λεπτό οι υπόλοιποι. Ζωηρό ενδιαφέρον, μακροσκελής κατάλογος των ομιλητών. Οι συντονιστές ήδη είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν την Υπουργό, οπότε παρακαλώ να μην ξεπεράσουν το δίλεπτο που δικαιούται ο καθένας. Ο κύριος ε, Ντές από το ΕΛΚ. Ο κύριος Ντέις του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι που έχουμε πάλι την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Αναφερθήκατε σε ορισμένα θέματα, θα προσπαθήσω να κρατήσω το πλαίσιο του χρόνου. Υπάρχει ανάγκη ανάληψης δράσεως για την ε, αξιορισμένων ανισορροπιών. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο και σας παρακαλώ και εσείς ως Προεδρία του Συμβουλίου να τα λάβετε υπόψη και να μας υποστηρίξετε. Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό εμπόριο, θα ήθελα να πω ότι στην Επιτροπή Γεωργίας παρα... το παρακολουθούμε και αποφασίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία να ζητήσουμε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την TTIP. Σημαντικό για τους γεωργούς μας είναι τα πρότυπα για την προστασία καταναλωτών ζώων και του περιβάλλοντος να διατηρηθούν. Αλλιώς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες. Μου είπαν άλλωστε σήμερα οι ε, εκπρόσωποι του γαλακτοκομικού μου συνεταιρισμού ότι ε, συμφώνησαν να εξαγάγουν 3.000 τόνους γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, κάτι το οποίο βεβαίως οφείλεται στο ότι διαθέτουμε συμφωνία με τη χώρα αυτή. Σε ό,τι αφορά το μέλλον τη γεωργική πολιτική, σα ζητώ την υποστήριξή σα Το Κοινοβούλιο έχει κάνει πολλέ προτάσει. Ο επίτροπο επίση, κατά τη γνώμη μου, δεν αρκεί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εκτελεστικές μονοπράξεις. Πρέπει να, αλλάξει, να αλλάξουν σε ορισμένα σημεία και οι κανονισμοί βάσεω σε συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα. Χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές που είναι αναγκαίες σε ό,τι αφορά την αστάθεια τιμών των γεωργικών προϊόντων και εδώ είναι ανάγκη να γίνουν αλλαγέ. Για παράδειγμα, το δυσκίνητο σύστημα παρεμβάσεων. Χρειαζόμαστε ένα ταχύτερο σύστημα που να επιτρέπει ταχύτερη αντίδραση. Λίγα ζητήματα που ήθελα να θίξω. Δεν βλέπω πουθενά χρονόμετρο, κύριε Πρόεδρε. Αλλά βεβαίω δεν θέλω να υπερβώ τον ε, χρόνο μου. Εύχομαι λοιπόν κύριε Υπουργέ σε εσά και στην Προεδρία σα καλή επιτυχία και εύχομαι να, η συνεργασία μας να είναι καρποφόρα. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα με το χρονόμετρο, αλλά εσείς τα καταφέρατε και τηρήσετε το χρόνο σας. Ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ να ευχηθώ καλή δουλειά στην κυρία Υπουργό Αναλαμβάνετε την Προεδρία του Συμβουλίου Γεωργίας σε εποχές δύσκολες για την Ευρώπη. Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για τον Brexit. Εποχές όπου παρατηρούνται εθνικιστικές ε, τάσεις, ε, ανησυχίες για το πεπρωμένο της Ευρώπης. Και παρόλα αυτά η Γεωργία αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα, μας προσφέρει παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Η κρίση του γάλακτος αποδεικνύει για άλλη μία φορά πόσο απαραίτητες είναι οι παρεμβάσεις ευρωπαϊκής κλίμακας, όπως είπατε και εσείς στην παρουσίασή σας. Τίθετο ζήτημα της αλληλεγγύης, διότι όλες οι χώρες ε, ε, πληρώνουν για τις χαμηλές τιμές του γάλακτος αλλά δεν ευθύνονται όλες για την τόσο υψηλή παραγωγή του γάλακτος στην Ευρώπη και τα εθνικά μέτρα δεν θα παραμείνουν αν ε, δεν έχουμε ευρωπαϊκά μέτρα θα συνεχίσουμε να έχουμε περισσεύματα Έχουμε το θέμα της Ρωσίας, το θέμα της γαλακτοσκόνης στην Κίνα. Εμείς παράγουμε γάλα γιατί δεν υπάρχει ακόμα απόφαση. Ε, δεν έχει βάλει τίποτα στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την Τρίτη στις 19 ο Επίτροπος Χόγκαν πρέπει να έρθει με σοβαρές ιδέες που να βάλουν σε κάποια πορεία την Ευρώπη. Γιατί αν η Ευρώπη δεν αποκριθεί, οι πολίτες μας δεν θα καταλάβουν τι κάνει αυτή η Ευρώπη. Συμφωνώ μαζί σας, είναι απαραίτητο να παρεύουμε για μια απλούστευση που να μην μειώσει τις παραβολωτικές προσπάθειες που έχουμε θελήσει σε αυτή τη νέα κοινή πολιτική και με τον greening. Αλλά το greening πρέπει να γίνει λιγότερο περίπλοκο τόσο για τους γεωργούς όσο και για τα κράτη-μέλη. Και οι δυνατότητες υπάρχουν. Αλλά χρειάζεται μια πρωτοβουλία ισχυρή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ και καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κούσμιουκ και δέκα δευτερόλεπτα πριν το πέρας του δίλεπτου και για να σας διευκολύνω θα σηκώνω το εργαλείο μου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Υπουργό για τόσο περιεκτική και ευρεία παρουσίαση των προθέσεων της Σλοβακικής Προεδρίας και χαίρομαι που αναλαμβάνει την Προεδρία μία χώρα από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, από αυτή την ομάδα των χωρών. Και καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τι προβλήματα έχετε στη Γεωργία, γιατί παρόμοια έχουμε όλες οι χώρες αυτής της περιοχής, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία έχουν παρόμοια προβλήματα στη γεωργία και έχουν πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές και έχουμε πληγεί ανεπανόρθωτα από το ρωσικό εμπάργο. Και επίσης ε, έχουμε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες στήριξης των γεωργών και χαμηλότερο επίπεδο άμεσων ενισχύσεων σε σχέση με τους γεωργούς των ε, δυτικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα ε, φλέγοντα τα προβλήματά μας και ελπίζω θα το λάβει υπόψη αυτό η Σλοβακική Προεδρία και θα πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, λάβει υπόψη στη λύση της τα ιδιαίτερα προβλήματα των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, πώς κρίνεται την επαναχώρηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την ε, επίλυση της κρίσης στην αγορά γάλακτος και στην αγορά οποροκυπευτικών. Δυστυχώ είναι ανεπαρκή η προτάση Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεδομένη τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζουν αυτοί οι κλάδοι. Επίση, τι γνώμη έχετε για τι διαπραγματεύσει ε, TTIP, τι συμφωνίε με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Θεωρείτε ότι η συμφωνία αυτή θα ευνοήσει ή θα απειλήσει την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέλλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Υπουργό που ήρθε και μας μίλησε στην Επιτροπή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία σας, γιατί έχετε πραγματικά μείζονες προκλήσεις να αντιμετωπίσετε. Αναφερθήκατε πολύ σωστά στην ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας στην κοινή γεωρική πολιτική. Και η δική μας Επιτροπή έχει υποβάλει σχετικές προτάσεις για τους ελέγχους, στην πολλαπλή συμμόρφωση. Υπάρχει έντονη ανάγκη απλούστευσης της γραφειοκρατίας. Αλλά εμείς κάνουμε το καθήκον μας, αλλά το Συμβούλιο δυστυχώς δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προτάσεις μας. Θα πρέπει να συμμετέχουμε πιο ενεργά και να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις μας. Σίγουρα χρειαζόμαστε κατεπηγόντω απλούστευση τη κοινή γεωρικής πολιτικής, ε, γιατί διαφορετικά αντιδρούν τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, οι πρακτικές μερικέ φορέ αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ ε, στην τροφική αλυσίδα, πολύ σημαντικό θέμα. Και η δασοκομεία, όπω είπατε. Γιατί μερικέ φορέ τα κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη. Έχουμε το Natura 2000 στην οδηγία για την προστασία του περιβάλλοντος και για 200 χρόνια είχαμε αρκετά βιώσιμη διαχείριση των δασών και μας ενοχλεί τώρα αυτή η παρέμβαση που διαπιστώνουμε. Γιατί πρόκειται για ένα αγαθό που μας ανήκει και είναι πολύ σημαντικό στις πολιτικές μας. Σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή εντοχή, θα πρέπει να φροντίσουμε να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όταν θεσμοθετούμε για τις ζωτροφές, για παράδειγμα. Είναι μεγάλο το φάσμα των δράσεων και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σένερα. Το χρονόμετρο λειτουργεί, παρακαλώ να το κοιτάζετε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Υπουργό και καλημέρα σας και πάλι. Θα ήθελα ε, για το Συμβούλιο της Δευτέρας ε, να σας ε, προτείνω στόχο να θέσετε επιτέλους ένα τέρμα στην πολιτική ουσιαστικά εκμυδένιση των αγορών. Θα συζητήσετε τη γαλακτοκομική κρίση. Θα ήθελα λοιπόν να σας παροτρύνω να μιλήσετε επιτέλους για μια δημόσια πολιτική, γιατί χρειαζόμαστε μια τέτοια δημόσια πολιτική για να μειώσουμε τη γαλακτοκομική παραγωγή στην Ευρώπη, να θεσπίσουμε μηχανισμούς ρύθμισης και να αρχίσουμε και πάλι να μιλάμε για μια τιμή που θα καλύπτει το κόστος παραγωγής και θα αμείβει τους παραγωγούς. Αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής γεωργίας και για το γαλακτοκομικό τομέα αλλά και για όλους τους τομείς παραγωγής. Γιατί σε τελική ανάλυση η κρίση που βιώνουμε οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε τόσο χαμηλές τιμές, τόσο τιμές κάτω του κόσμου που δεν μας επιτρέπουν να, επιβιώνουμε και να βιοποριζόμαστε. Και παραλαμβάνω, αυτό το θέμα αφορά όχι μόνο το γαλακτοκομικό τομέα, αλλά και τους άλλους ε, γεωργικούς κλάδους. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά και τη ΤΥΠ με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα ήθελα να επισημάνω δύο τινά. Ναι. Θα ήθελα ε, να συμπεριλάβετε στη συζήτηση και το ζήτημα της μη επικύρωσης της ΕΤΑ, γιατί είναι αντιδημοκρατική συμφωνία, πολύ επιθετική και πολύ επιζήμια για τους Ευρωπαίους Γεωργούς. Και θα ήθελα για τους ίδιους λόγους να διακόψετε και τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το TTIP. Και μια και ο χρόνος μου εξαντλείται, θα ήθελα να σας υποβάλω και μια ερώτηση. Είπατε ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να είναι ελκυστική για τη γεωργία. Συμφωνώ. Ε, όχι μόνο για του τωρινού γεωργού, αλλά και για τι επερχόμενε γενιέ. Συμφωνώ. Μιλήσατε όμω ότι θα πρέπει, ε, είπατε, θα πρέπει να είναι ελκυστική και για του επενδυτέ. Τι εννοείτε, σε ποιου ε, επενδυτέ αναφέρεστε και θα πρέπει, θα πρέπει κάτι τέτοιο να είναι συμβατό και με τι ανάγκε και τα συμφέροντα των γεωργών τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Χόισλινγκ. Ναι, καλώ ορίστε και από εμάς και τι καλύτερε ευχές μας ε, για την Προεδρία του Συμβουλίου. Εύχομαι, ελπίζω μάλλον αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία που είπατε ότι είναι η βιολογική γεωργία να προωθηθεί επαρκώ ε, και ελπίζουμε ότι στο τέλο τη Προεδρία σα θα έχουμε τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου στο Κοινοβούλιο είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να κάνουμε συμβασμούς. Ε, χθες ε, μιλήσαμε με τον Επίτροπο και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Αλλά βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές, σε μια δύσκολη κατάσταση όπου η Προεδρία του Συμβουλίου ελπίζω να συνεχίσει να παίρνει αποφάσεις, να παίρνει και αποφάσεις για το τομέα των γαλακτοκομικών δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης. Όχι απλά να σημειώνεται τι συμβαίνει, αλλά να βοηθήσετε να επανέλθει η ισορροπία της αγοράς μακροπρόθεσμα. Δεν θα τα καταφέρουμε αν δεν καταφέρουμε η προσφορά να συμβαδίζει με τη ζήτηση. Δεν είναι απλά θέμα του να, το, να σημειώνουμε που βρίσκονται οι αγορές. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε ορισμένους κανονισμούς της αγοράς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλή ιδέα βέβαια, αλλά την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε κάποιες σαφείς ενδείξεις, τις οποίες χρειάζονται οι αγρότες για να εργαστούν. Αλλιώ οδεύουμε προς την καταστροφή. Αντίθετα με του συναδέλφου μου όσον αφορά τις επικρίσεις κατά του TTIP και του ΣΥΤΑ, δεν θεωρούμε ότι απλά είναι ένα θέατρο. Θεωρούμε ότι οι γεωργοί της Ευρώπης θα χάσουν μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις και πρέπει να υπερασπίσουμε σοβαρά τα συμφέροντά τους. Ελπίζω λοιπόν ότι ο Επίτροπος θα αντιληφθεί ότι οι ελεύθερες συναλλαγές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να πραγματοποιούνται θυσιάζοντας τη Γεωργία. Οι, τα συμφέροντα των γεωργών μας πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε άλλους να τους ελέγχουν και να ε, λένε προχωράτε με απελευθέρωση των αγορών χωρίς κανένα όριο. Και κάτι άλλο ακόμα. Ξέρω ότι τονίσατε τη σπουδαιότητα των κτηνιατρικών φαρμάκων που χρειάζονται κάποια πρόοδο. Είναι σημαντικό. Και η χρήση των αντιβιωτικών αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι των όσων πρέπει να αλλάξουμε. Σα εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία με αυτή τη δέσμη μέτρων για τα κτηνιατρικά φάρμακα για τη βελτίωση τη υγεία των ζώων. Ευχαριστώ. Thank you, Well, good morning, I'm sorry. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Έχασα το πρωινό, συγγνώμη, ήταν απόφευκτο για μένα. Ως Βρετανός βουλευτής με απασχολούν λιγότερο οι μακροπρόθεσμες πτυχές ε, της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής φυσικά, αλλά υπάρχουν κάποιες βραχυπρόθεσμες πτυχές με απασχολούν και η πρώτη είναι αυτή η πρόσφατη στάση του Συμβουλίου που υφίσταται άνετα από τα πράσινα λόμπι ε, εκβιασμούς όσον αφορά τα φυτοφάρμακα και αυτό με ανησυχεί. Εσείς ε, θα ήσασταν, πρέπει να ήσασταν στο Συμβούλιο όταν ε, δεν ενέκριναν το γλυφοσάτ, ε, τη γλυφοσάτη για τα επόμενα χρόνια θα έρθουν και συζητήσει και για άλλα φυτοφάρμακα μέσα στους επόμενους μήνες που θα απαγορευτούν λόγω της πίσης του πράσινου λόμπι. Και αυτό είναι πολύ ενσχετικό πιστεύω. Μετά αναφέρατε τη βιολογική γεωργία, κανόνες που μπορεί να επηρεάσουν εμάς στη Βρετανία. υπάρχουν ε, δύο αντιφάσει αυτά που είπατε. Από τη μια λέτε περισσότεροι κανόνε στη βιολογική γεωργία θα την καταστήσουν πιο ανταγωνιστική. Ε, με ένα εντύπωση μου είναι ότι θα γίνει λιγότερο ανταγωνιστική. Το άλλο, η άλλη αντίφαση είναι αν θέλετε να είναι εμβληματική πρωτοβουλία, εμβληματική πολιτική ή βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θεωρώ περίεργο. Αυτό αντίκειται με το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αλλάξει τον καιρό στον κόσμο αν είναι να πάμε στην βιολογική καλλιεργία, πρέπει να καλλιεργούμε, να καλλιεργούμε και να καλλιεργούμε. Επειδή δεν θα χρησιμοποιούμε λιπάσματα το οποίο σημαίνει θα καλλιεργούμε μεγαλύτερε εκτάσει, εκλείοντα ε, διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο είναι ο δημόσιο εχθρό αριθμό 1. Λοιπόν, θα σταματήσω τώρα ε, πριν να αρχίσει να σηκώνει το χέρι του και σε χτυπήσει κατά λάθο ο κύριο Πρόεδρο. Τι θα κάνουμε χωρί αυτόν. Σας ευχαριστούμε Βέβαια, η σύγκριση παρά ήταν ε, τραβηγμένη. Ο κύριος Λοζό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την επίσκεψη, κύριε Υπουργέ. Έχετε πολύ, πολλά ψωμιά να φάτε. Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Και ξέρετε τι προβλήματα έχουμε και στη Γαλλία σε όλες τις παραγωγές. Ε, απορροκυπευτικά, γάλα, κτηνοτροφία, ακόμη και στα δημητριακά. Και οι καλλιεργητές σιτηρών υποφέρουν σήμερα στη Γαλλία εξαιτία τη κακοκαιρία των αντίξεων καιρικών συνθήκων. Ειδικά στην κεντρική Γαλλία είχαμε φοβερή κακοκαιρία και μερικοί γεωργοί λόγω των πλημμυρών έχασαν τελείω την παραγωγή τους. Καταστράφηκαν οι σοδιές τους. Έχουμε σημαντική μείωση παραγωγή, η, η παραγωγη που μας έχει απομείνει δεν είναι ιδιαίτερα ποιοτική. Έχουμε το πρόβλημα με τις ενισχύσεις, το ρωσικό εμπάργο, τη επερχόμενη διατλαντική συμφωνία που απειλεί να καταστρέψει τους γεωργούς. Στη Γαλλία είχαμε πάνω από 600 αυτοκτονίες γεωργών τραγικά γεγονότα, ιδιαίτερα ανησυχητικά. 14% των Γάλλων γεωργών δήλωσαν ε, κατά την αρχή του έτους ότι θα διακόψουν τις γεωργικές δραστηριότητες. Σήμερα έχει ανέβει το ποσοστό. Μερικοί μιλούν για 20-25% των Γάλλων γεωργών που από φέτος ε, θα σταματήσουν τη δραστηριότητά τους. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να βοηθήσετε τους γεωργούς προκειμένου να ξεπεράσουν αυτή την τραγική κατάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στις ε, μονόλεπτες παρεμβάσεις των λοιπόν μελών της Επιτροπής Γεωργίας. κυρία Κέστιγκερ, για ένα λεπτό. κυρία Κέστιγκερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Υπουργέ. Το βρίσκω ιδιαίτερα ε, σημαντικό ότι έχετε λάβει ως κέντρο ε, βάρος της πολιτικής σας και την δασοκομεία. Ειδικά σε αυτό το εξάμεινο αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέε προτάσει, οι οποίε θα έχουν σημαντικέ επιπτώσει στην Ευρωπαϊκή Δασοκομεία. Επιθυμώ να επαναλάβω ότι ιδίω για το non-ETS και για το LULUCF μας ενδιαφέρει να γίνει σαφής η διάκριση ανάμεσα στο πράσινο ε, διοξείδιο του άνθρακος το οποίο προέρχεται από την αναπνοή των φυτών και αυτό που προέρχεται από το έδαφος και που εν τέλει παραμένει εκεί. Πολύ συχνά λείπει αυτή η διάκριση παρόλο που ε, σε αυτήν εγκύπτουν πολλοί εμπειρογνώμονες. Στα πλαίσια της Προεδρίας σας θα σας παρακαλέσω λοιπόν σε όλες τις σχεδιαζόμενες ε, συζητήσεις να το λάβετε υπόψη, καθώς και για το κριτήριο βιωσιμότητας για την βιομάζα. Να φροντίσετε δηλαδή να γίνεται καθαρά η διάκριση αυτή, διότι αλλιώς δεν εξυπηρετούμε την δασοκομεία. Ε, σας παρακαλώ επίσης, όταν θα εφαρμόσετε την στρατηγική για τη δασοκομεία, να μην χάσετε από τα μάτια και την ανάγκη αναβάθμισης της Επιτροπής Δασοκομείας. Το έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προβλέψει δηλαδή μέτρα εφαρμογής και σας παρακαλώ και στα πλαίσια της επικουρικότητας να φροντίσετε για την εφαρμογή της στρατηγικής δασοκομείας. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό έχετε ο καθένα παρακαλώ, μην το ξεπερνάτε. Κυρία Γκαρσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Υπουργό που ήρθε. Μου είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, τις καταχρήσεις που γίνονται στην τροφική αλυσίδα και είπατε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους γεωργού. Ερωτώ λοιπόν, θα στηρίξετε την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, θέσπιση σχετικής ε, νομοθετικής διάταξης και τι θα κάνετε προκειμένου να έχουμε επιτέλους ε, νομοθετικές διατάξεις που θα διέπουν την τροφική αλυσίδα. Την επόμενη εβδομάδα στη, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας θα εξετάσετε έκτακτα μέτρα για το γάλα. Συμφωνείτε με τη θέση της Γαλλίας, Ισπανίας και άλλων χωρών που ζητούν αύξηση των τεμήνιμης ενισχύσεων, το διπλασιασμό των ενισχύσεων αυτών μάλιστα γιατί όλα αυτά θα είναι νέα μέτρα για τον έλεγχο τη γαλακτοκομική παραγωγή. Συμφωνείτε ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα του γάλακτο θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε άλλου ε, γεωργικού τομεί, όπω τον τομέα των αποκυπευτικών που επίση ταλανίζονται από την κρίση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Αγγιλέρα, αντιπρόεδρός μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Χθες είχα την ευκαιρία να παραστώ στο πρόγευμα των συντονιστών μαζί σας, ε, των συντονιστών της Γεωργίας και των συντονιστών της Επιτροπής Αλίας. Εργαστήκαμε πολύ εντατικά αυτό το διήμερο. Θα σας αναφέρω ένα θέμα φλέγων. Τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την κρίση και τα έκτακτα μέτρα που θα εξετάσετε στο επόμενο Συμβούλιο. Τα μέτρα του Σεπτεμβρίου ε, για την αντιμετώπιση κρίσης ε, δυστυχώς ε, απέβησαν αναποτελεσματικά και ανεπαρκή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε τέτοιου τους μέτρα, αλλά να λάβουμε υπόψη πραγματικές ανάγκες της γεωργίας. Η τροφική αλυσίδα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν κάποιες αποφάσεις πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, γιατί τα εθνικά μέτρα για την τροφική αλυσίδα είναι επίσης άχρηστα. Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι είναι αναγκαία η αμοιβαιότητα σε αυτές τις συμφωνίες. Θα πρέπει να πετούμε την αμοιβαιότητα σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτουμε με τρίτες χώρες. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι είμαι η συγγήτρια της έκθεσης για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Η συζήτηση ήδη έχει γίνει και στη δική μας επιτροπή και στην ΕΜΒΗ για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Ελπίζω ότι θα προωθηθούν και τα δύο θέματα κατά τη διάρκεια τη Σλοβακική Προεδρία. Ευχαριστώ. Κύριος Νταντάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον ακούσαμε τα όσα είπατε. Το λέω και εκ μέρους του συνάδελφου Μαγκίνες, ε, της συνάδελφου Μαγκίνες που ζητά συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ σήμερα το πρωί. Ακούσαμε με πολύ προσοχή λοιπόν ε, τα όσα είπατε για τη λειτουργία της ε, τροφικής αλυσίδας. Δυστυχώς το, ε, το, ε, το ψήφισμα που ψηφίσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο πριν λίγες εβδομάδες είναι ισχυρό. Θα ήθελα πέραν της απλής λειτουργίας της τροφικής αλυσίδας να κάνω μια προσθήκη. Πιστεύω ότι στο Συμβουλίο Υπουργών πρέπει να φροντίσετε για την εφαρμογή των άρθρων της συνθήκης που, αφορά το δικαίωμα ανταγωνισμού όπως εφαρμοστεί στη Γεωργία γιατί από τη μια απόφαση μέχρι την άλλη τελικά αυτή η αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη και η Κομισιόν συνέχεια πάει να μας πάει προς το γενικό καθεστώς. Η Γεωργία έχει κάποιε ιδιαιτερότητες τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε και να αξιοποιούμε σε όλα τα, στις φάσεις της αλυσίδας. Δύο άλλα σημεία που ήθελα να αναφέρω όσον αφορά την κατάσταση των αγορών. Σας εύχομαι ένα πράγμα κύριε Υπουργέ, να δώσετε κάποια επιθυμία για Ευρώπη στους υπουργούς μας ξανά, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι στο Συμβούλιο δεν θέλει κανείς πλέον πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική. Ο καθένας το δικό του χωράφι υπερασπίζεται. Εμείς ούτως πράγμα στο Κοινοβούλιο, θέλουμε το ίδιο και στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριο Σμάτο Αντρόβερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Η γεωρική κρίση είναι πια κάτι το προφανέ και θα κληθείτε να την αντιμετωπίσετε και εσεί στην Προεδρία σα. Αλλά είναι ακόμη πιο προφανή και έκδηλη αυτή η κρίση στι εξόχω απόκεντρε ε, περιοχέ. Στα Κανάρια, για παράδειγμα, τα οποία κατάγομαι. Το ΠΟΣΕΙ είναι ένα μηχανισμό, ε, δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη, είναι απαραίτητο μηχανισμό για τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Και κατά τη διάρκεια τη Σλοβακικής Προεδρία ε, θα γίνει αναθεώρηση του ΠΟΣΕΙ ε, θα πρέπει να το προσέξετε ιδιαίτερως γιατί είναι μεγάλο το διακύβευμα. Σε ό,τι αφορά τι εμπορικέ συμφωνίε, δύσκολη η εξέβρεση ισορροπία μεταξύ διεθνούς εμπορίου και Γεωργία. και πολύ φοβάμαι ότι πολλέ φορέ την ύφη και τα σπασμένα την πληρώνουν οι γεωργίε στις εμπορικέ συμφωνίες. Το ίδιο μάλιστα μάλλον θα συμβεί και με το Εκουαδόρ και με προβληματίζει η κατάσταση των παρανοπαραγωγών στη Γεωργία. Είχαμε τεράστια προβλήματα με τι ντομάτες και τη σχετική συμφωνία με το Μαρόκο. Φοβάμαι ότι ίδια προβλήματα θα έχουμε και με το TTIP. Επίσης, αμοιβαιότητα είναι απαραίτητο να το διεκδικούμε, γιατί πολύ φοβάμαι ότι οι καλλιεργητές τρίτων χωρών θα χρησιμοποιούν απαγορευμένες τροφές και παρόλα αυτά εμείς θα εισάγουμε προϊόντα από αυτές, ενώ απαγορεύουμε στους δικούς μας γεωργούς στα Κανάρια, για παράδειγμα, στη Μαδέρα να χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες. Ευχαριστώ. Κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλύψατε μεγάλο φάσμα στα, με τα εισαγωγικά σας λόγια. Όμως υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ επίγοντα, δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο. Το πιο επίγον σήμερα είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουν επαρκές εισόδημα οι αγρότες, τουλάχιστον να μπορούν να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και ένα ελάχιστο κέρδος, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν Το εισόδημα των γεωργών είναι βεβαίως το εισόδημά τους από την ε, παραγωγή που πωλείται καθώς και κάποιες πρημοδοτήσεις ή κάποιες ε, ενισχύσεις. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις άμεσες ενισχύσεις που λαμβάνουν οι ε, αγρότες στις διάφορες χωρισμένοι. Μήπως πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί και να ευθυγραμμιστεί. Ευχαριστώ κύριο Σερεμπέγκα. Ε, Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, η Σλοβακία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στιγμές βαθιάς κρίσης. Και δεν είναι μονάχα μια κρίση. Πολλές κρίσεις που μας απασχολούν βαθύτατα και μιλώ για την κρίση του προσφυγικού που θεωρώ είναι, ότι είναι από τα σημαντικότερα, τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και μάλιστα για τις τελευταίες δεκαετίες. Τα δύο τελευταία χρόνια χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διοχετεύσει σημαντικά κονδύλια από τον προπολογισμό για να διευκολύνει την επίλυση της κρίσης αυτής. Η λύση που σκέπτονται ορισμένοι είναι να τροποποιήσουν την ε, τον προορισμό κάποιων κονδυλίων από την γεωργία και να τα διοχετεύσουν στο προσφυγικό. Δεν νομίζετε ότι αυτό θα οδηγήσει σε έλλειψη ισορροπίας της αγροτικής οικονομίας. Ευχαριστώ κυρία Νόιχλ. Μετά από τον προλαλήσαντα, τι να πω, ε, να, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η τροπή που έδωσε. Χαίρομαι που σας γνωρίζω κύριε Υπουργέ. Συγκεκριμένη παράκληση. Παράκληση να χορηγήσετε βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε να καταθέσει μελέτη για τις σορευτικές επιπτώσεις των συμφωνιών ΣΕΤΑ, ΤΙΤΙΠΗ και ΜΕΡΚΟΣΟΥΡ. Εάν δηλαδή ισχύσουν και οι τρεις αυτές συμφωνίες, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Όχι δηλαδή κάθε μια συμφωνία ξεχωριστά, αλλά το σύνολο των ε, συμφωνιών αυτών ποιε επιπτώσει θα έχουν στην Ευρώπη. Βεβαίω οι χώρε Μερκοσούρ επιθυμούν να εξαγάγουν στην Ευρώπη προϊόντα τα οποία είναι ε, του ενδιαφέροντος και των άλλων συμφωνιών. Ακόμα δεν έχει κατατεθεί η μελέτη αυτή. Πριν νομίζω να υπογραφτεί έστω και μια από τις συμφωνίες αυτές πρέπει να ξεκαθαριστεί η εικόνα τι θα γίνει εάν βάλουν το πόδι στην αφετηρία και οι τρεις αυτές συμφωνίες. Γι' αυτό σας παρακαλώ στη διάρκεια της Προεδρίας σας, πολύ συγκεκριμένα, να φροντίσετε να διαβαστεί η μελέτη αυτή στις χώρες μέλη και βέβαια και στους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τις ευχές μου στην Προεδρία. Τέσσερα σχόλια. Πρώτο, για τις αθέμητες πρακτικές στην την τροφική αλυσίδα. Σημαντικό αυτό είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεύτερο, τρίτο, η όλο και αυξανόμενη συμβασία της δασοκομείας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επειδή 8% παγκοσμίω των ε, εκπομπών ε, οξυδιών του άνθρακα είναι, προέρχεται από την παραγωγή τσιμέντου, να αντικαταστήσουμε το τσιμέντο με ξύλο στις κατασκευές, στις οικοδομές. Το ίδιο για την χαλιβουργία βεβαίω και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύλο με ειδικού τρόπους που είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και τέλο, μην αγνοείτε πόσο προβληματικέ είναι κάποιε γεωργικές πολιτικέ που ακολουθούνται τώρα για την αλλαγή του κλίματο. Όμω, από την άλλη μεριά, εάν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, η γεωργία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Άκουσα με προσοχή τα όσα είπατε για την ανανέωση της γεωργίας. Ποιες είναι οι προθέσεις σας όσον αφορά την επόμενη ε, κοινή γεωργική πολιτική με οριζόντα το 2020 σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό πλαίσιο πώς θα καταφέρουμε να έχουμε μια οικονομικά βιώσιμη, περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργία που θα διασφαλίζει την ασφάλεια, την γεωργική αυτονομία και το γεωργικό μοντέλο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Μιλήσατε για ε, τα διοικητικά θέματα. Πιστεύω ότι το σημαντικό είναι να σταθεροποιήσουμε τους όλους κανονισμούς που υπάρχουν. Ε, αναφέρθηκε το ζήτημα των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Ε, πρέπει να δούμε ποιες θα είναι, τι θα γίνει και με τι ποσοστώσει μάλιστα του Βόλου Κρέατο ε, με τη Μεγάλη Βρετανία. Ο κύριο Άντριου. Α, ο κύριος Άντριου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Υπουργό. Να συμπληρώσω κάτι στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα για την κρίση, όπω επισημάνεται, ειδικότερα για το γάλα. Είστε επίσημα διατεθειμένοι να υλοποιήσετε το άρθρο 122 του της κοινή αγοράς. Ε, δεύτερον, ε, να ρωτήσω κάτι για την ε, βιολογική γεωργία. Προβλέπετε επίσημα να οριστεί ολοκληρωθεί αυτός ο φάκελος πριν το τέλος της Σλοβακικής Προεδρίας που ξεκίνησε με την Ολλανδική Προεδρία. Τώρα για τη ΣΕΤΑ είπε και η συνάρφος Ντελαέ, συμφωνώ και εγώ, το ζήτημα του κινδύνου είναι πολύ σημαντικό για το βόλιο κρέας θα πρέπει να προσέχουμε διότι η ειδικευμένη παραγωγή ε, δεν έχει την ίδια διαδρομή από ό,τι γνωρίζουμε για τα εγωπρόβατα. Έχετε λοιπόν υπολογίσει τον κίνδυνο αυτού που ενέχει αυτός ο τομέας. Ευχαριστώ και σας κύριε Πρόεδρε και σας κύριε Υπουργέ. Πολλά λέχθηκαν ήδη για το γάλα. Επιθυμώ να τονίσω ίσως και με αριθμούς, ότι το 2015 πάνω από 3,5 εκατομμύρια τόνοι έλειπαν από την ε, αγορά μας. Επαναλαμβάνω την ε, ερώτηση και άλλων συναδέλφων. Αν είστε διατεθειμένοι να προωθήσετε μια μείωση των, ποσών, των, ποσο, ε, παγωμένων ποσών στην Ευρώπη. Άλλο θέμα τώρα. Λοιπάσματα. Καινοτομίε. Θέλω να μάθω πιο συγκεκριμένα ποιε δυνατότητε καινοτομία βλέπετε. Ιδίω για, για τα ψυχανθή. Ο κύριος Σάντος. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία. Γιατί όσο πιο επιτυχημένη η Προεδρία, τόσο τις επιτυχίες θα τις νιώσουμε όλοι στη Γεωργία. Ε, χαίρομαι που έχετε ως προτεραιότητα να υιοθετήσετε συγκεκριμένα μέτρα για να εξορροπήσετε τη θέση των γεωργών στην τροφική αλυσίδα και στην αλυσίδα αξιών. Γιατί οι γεωργοί αξίζουν μια αξιοπρεπή τιμή για το έργο τους. Και δυστυχώς οι χαμηλές τιμές πλήττουν κυρίως ε, τους γεωργούς και οι χαμηλές τιμές και οι μεγάλες χρήσεις των μεγάλων σούπερ μάρκετ και οι μονομερείς μερικές φορές ε, συνθήκες και όροι που τους επιβάλλονται στις συμβάσεις. Επίσης ε, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την κατάσταση της γαλακτοκομικής παραγωγής στην Ευρώπη. Εγώ κατάγομαι τις Αζόρες, μια εξόχως απόκεντρη περιοχή που παράγει το 30% του πορτογαλικού γάλακτος και η τοπική οικονομία εξαρτάται ιδιαίτερως από τη γεωργία και ιδιαίτερα τη γαλακτοκομική παραγωγή. Δυστυχώς με την κρίση έχει πληγεί ο κλάδος που πασχίζει ε, να παράγει ποιοτικό γάλα εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες ε, ε, Δυστυχώ υπάρχουν μεγάλε γεωγραφικέ ανισορροπίε. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα προσπίζει όλου του γεωργού και όχι μερικού μόνο. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ιδιαίτερε ε, και κατάλληλε προτάσει. Και θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. Και περιμένουμε ιδιαίτερες ιδιαίτερε προσδοκίε ε, και αδημονία το επόμενο Γεωργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Σα ευχαριστώ, κύριο Φλάνεγκαν. Ευχαριστώ πολύ η δουλειά σας φυσικά τώρα δεν απλά να εκπροσωπείτε τους γεωργούς από τη χώρα σας, αλλά τους γεωργούς όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ότι έχει μείνει μετά από το Brexit. Και αναρωτιέμαι τώρα, τι κατεύθυνση θα ακολουθήσετε όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όσον αφορά την πρόσβαση των Ιρλανδών γεωργών στην Βρετανική αγορά και αντιστρόφως δεδομένου ότι η Ιρλανδία βρίσκεται σε μια πολύ ξεχωριστή θέση εδώ, σε δύσκολη θέση, όπου ξαφνικά θα έχουμε χερσαία σύνορα με ουσιαστικά μια χώρα που θα βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναρωτιέμαι η δική σας θέση ποια θα είναι. Θα υπερασπίστε τα συμφέροντα όλων των γεωργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θα λάβετε υπόψη και τα συμφέροντα της Ιρλανδίας ή θα ακολουθήσετε την πορεία ότι οποιοδήποτε φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τον μαλώσουμε, να τον τιμωρήσουμε ώστε να μην το ξανακάνει κανένας. Ελπίζω λοιπόν να δείξετε αλληλεγγύη σε άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν περιμένω και πολλά θετικά. Ευχαριστώ κύριε Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Θεωρώ ότι επιλέξατε με μαεστρία τις προτεραιότητες προεδρίες Αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές είναι η πληγή και ο καρκίνος της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Επίσης η ανάγκη να προστατεύσετε τα δάση δίνεται προτεραιότητα στην δασοκομεία. Είναι σημαντικός παράγοντας προστασίας του περιβάλλοντος με τη δέσμευση του άνθρακα που πραγματοποιούν. Επίσης ε, ε, θα ήθελα να ε, καλωσορίσω και εκπροσώπους της ε, Κροατικής Γεωργίας που περιμένουμε ανυπομονησία τις απαντήσεις Επίσης, μιλήσατε για την κρίση στη Γεωργία και τις θεομηνίες και την κακοκαιρία που την πλήττουν. Για παράδειγμα, τον ε, Απρίλιο είχαμε τεράστιες ζημιές από κακοκαιρία στην Αυστρία, Κροατία, Σλοβενία, Ρουμανία και έχουν υπολογιστεί οι ζημιές στο 1 δισεκατομμύρια, Έχουν καταστραφεί δάση, η αμπελουργία μας ε, και άλλες γεωρικές παραγωγές. Είχαμε την κρίση που ξεκίνησε και με το, από το ρωσικό εμπάργο, Έχουμε τις κακοκαιρίες, τις θεομηνίες. Δεν πιστεύετε ότι πέραν του γεωρικού προϋπολογισμού θα μπορούσαμε να συστήσουμε και ένα έκτακτο ταμείο αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών για να βοηθήσουμε τους γεωργούς μας. Ευχαριστώ. Κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη εργασία σας. Με ενδιαφέρει η ενιαία αγορά. Εκεί αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι το ρωσικό εμπάργκο έπληξε την ευρωπαϊκή αγορά αγροτικών προϊόντων. Πολλές χώρες μέλη και πολλούς αγρότες που είχαν μάλιστα άμεσες σχέσεις με τη ρωσική αγορά. Αυτοί αποζημιώθηκαν εν μέρη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι καλό. Όμως τα προϊόντα των αγροτών αυτών διοχετεύτηκαν σε χώρες που δεν είχαν άμεσες σχέσεις με τη ρωσική αγορά και αυτό έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Στη Ρουμανία για παράδειγμα πωλείται γάλα κάτω από 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο. Είναι αλήθεια κύριε Υπουργέ και μπορείτε να το ελέγξετε. Και γνωρίζουμε ότι το κόστος παραγωγής του λίτρου γάλακτος είναι 18 λεπτά του ευρώ. Χοιρινό πωλείται 80 λεπτά το κιλό, ενώ το είναι πάνω από 1 και 20 το κόστος παραγωγής. Ο κύριος Νίκολσον, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα συμφωνώ με τον κύριο Νταντέν. Τονίζει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εσείς καλά αρχίσατε. Η αγροτική οικονομία σας χρειάζεται. Συνεχίστε λοιπόν με τον ίδιο ρυθμό. Ερώτηση. Προβλέπετε εννέα τριμερείς διαλόγους ή μάλλον έχουν ήδη γίνει εννέα τριμερείς διαλόγοι για τα βιολογικά προϊόντα υπό δύο διαδοχικές προεδρίες. Η δική σας προεδρία πώς θα σπάσει το αδιέξοδο στον φάκελο αυτό. Θα ζητήσετε αναθεωρημένη εντολή. Αυτό δεν πάει πουθενά κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν το ξεχνούμε. Και εσείς κύριε Φλάνναγκαν. το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμα εγκαταλείψει την Ευρώπη. It, means some haven't jumped the ship yet. Σημαίνει ότι κάποιο δεν έχει πηδήξει ακόμα από το πλοίο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ κύριε Σφερά. Κύριε Υπουργέ, το κακό στην Ευρώπη είναι ο υπερβολικός νεοφιλελευθερισμός. Πρέπει να σταματήσουμε τις συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών που θα καταστρέψουν τις κτηνοτροφίες μας, την κτηνοτροφία μας και τους γεωργούς μας. Αυτές οι συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών θα οδηγήσουν σε κακής ποιότητα προϊόντα, θα καταστρέψουν τις ε, ε, ονομασίε προέλευσή μα. Πρέπει να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή κληρονομιά, η οποία βρίσκεται υπό απειλή από όλε αυτέ ε, τι ολέθριε συνθήκε. Είναι η γεωργία και η γη μα ε, ε, μια κληρονομιά της οποίας κληρονόμοι είμαστε εμείς και πρέπει να την υπερασπίσουμε, να την προστατέψουμε. Αλλιώς οι άλλες χώρες όπως το Ενωμένο Βασίλειο θα φύγουν και θα έχουν δίκιο. Αυτό το θέμα παίρνει αρκετή συζήτηση. Η κυρία Μόη. Ε, κυρία Υπουργέ, αξιότιμη συναδελφή. έχει ξεκινήσει ήδη η Σλοβική Προεδρία της εργασίας της για ένα εξάμενο το οποίο θα είναι ε, γεμάτο γεγονότα. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η διαπραγματεύση για συνθήκες με τη ΣΥΠΑ, τον Καναδά και την Κίνα η Ευρώπη. Δεδομένων αυτών των συμφωνιών, θέλω να επιθυμίσω στην Προεδρία μία από τις βασικές προτεραιότητες, όπως θεωρώ εγώ, για την Επιτροπή αυτή. Αναφέρομαι στο φάκελο για το cloning food, όπου είμαι και εγώ συνεισηγήτρια και για το οποίο έχει δώσει ήδη την του το Κοινοβούλιο. Από τη στιγμή που εδώ το ζήτημα είναι η προστασία της υγείας και της διατροφικής ασφάλειας των πολιτών μας και της καλής ευημερίας των ζώων, πρέπει οπωσδήποτε το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσει ένας τριμερής διάλογος, ώστε να συνεχιστεί η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία. Αυτό θα έδινε ένα σημαντικό μήνυμα από τη νέα Προεδρία. Ε, θέλουμε να δραστηριοποιηθεί για αυτό το σημείο, ώστε όλες οι νομοθεσίες να ολοκληρωθούν υπό τη δική σας εντολή. Λοιπόν, σας παροτρύνω να λάβετε υπόψη τα αιτήματά μου και με την ευκαιρία σας εύχομαι καλή, καλές εργασίες. Σας ευχαριστώ. Περίπου 30 ευρωβουλευτές έλαβαν το λόγο στη συζήτηση. Ήρθε η ώρα σας τώρα κύριε Υπουργέ. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι στις 10.30 ε, έχετε και συνέντευξη τύπου. Οπότε έχετε το λόγο και περιμένουμε τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Ε, και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Η πιο συχνό, συχνότερη ερώτησή σας έχει σχέση με την κατάσταση στην αγορά και ιδίω στην αγορά γαλακτοκομικών από τους κύριους Τεκάστρο, Κόσμιν, Ροντρίγκε και από πολλούς άλλους εκ των συναδελφών σας. Η κατάσταση στην αγορά είναι πράγματι κρίσιμη και δεν είμαι βέβαια υπουργό Γεωργίας για πολύ μεγάλο διάστημα. Έχω συμμετάσχει σε συναντήσεις που πάντοτε περίχαν στην ημερήσια διάταξή τους και αυτή την κρίση στην αγορά. Δύσκολη κατάσταση η οποία χρειάζεται αποτελεσματικές λύσεις και όσο χρόνο χάνουμε με αδράνεια τόσο, περισσότερο, τόσο περισσότεροι γεωργοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις αγροτικές τους δραστηριότητες. Ε, μιλήσατε εσείς για γεωργούς στην ε, Γαλλία, στη Σλοβακία και αλλού. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ισορροπούν ζήτηση και αγορά στην αγορά γεωργικών προϊόντων και αυτό προκαλεί τα προβλήματα. Τώρα προετοιμαζόμαστε για το Συμβούλιο του Ιουλίου όπου αναμένεται να ληφθούν πολλά μέτρα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να προπαρασκευάζουμε την λήψη μέτρων για τις επόμενες ε, διασκέψεις του Συμβουλίου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προπαρασκευάζουμε κοινή συνεδρίαση της High Level Group τον Σεπτέμβριο της Task Force για τα γαλακτοκομικά και θα συντάξουμε έκθεση για την δέσμη μέτρων για τα γαλακτοκομικά. Υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναζητεί νέες δυνατότητες εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων των Ευρωπαίων γεωργών και τρόπους να αντιμετωπιστεί η κρίση στον ε, τομέα αυτό. Στις 16 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί διάσκεψη υψηλού επίπεδου για το γάλα και τα γαλακτοκομικά, όπου θα παρουσιάσουμε εμείς μακροπρόθεσμες λύσεις, διότι η γαλακτοκομική κρίση δεν χρειάζεται μόνο βραχυπρόθεσμες λύσεις, χρειάζεται ιδίω μακροπρόθεσμες λύσεις για να στεθεροποιηθεί η κατάστασή της στο μέλλον. Θα προσπαθήσουμε θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και θα προπαρασκευάσουμε κάθε δυνατό μέτρο για να σταθεροποιήσουμε την αγορά και να συμβάλλουμε σε μια σταθερή και δίκαιη αντιμετώπιση των γεωργών μέσα στην τροφική αλυσίδα. Εφόσον μπορέσουμε να κατανείμουμε σωστά τα περιθώρια κέρδους, αυτό θα επιτρέψει να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των γεωργών και να εξασφαλιστούν και μελλοντικέ γενναίες στην γεωργία τα πάντα αλληλοσυνδέονται και η ίδια η κρίση είναι από τις προτεραιότητες, είναι η προτεραιότητα της Σλοβακικής Προεδρίας για να βελτιώσουμε, όπως είπα, την θέση των αγροτών στην τροφική αλυσίδα. Σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα που σας απασχολούν, όπως τα οποροκυπευτικά ο τομέας των απορροκυπευτικών. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του τομέα αυτού. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο εκεί, μα δεν μόνο στα γαλακτοκομικά η κρίση, αλλά και στα απορροκυπευτικά. Αναζητούμε λύσεις και εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποσχεθεί ότι θα επαναεξετάσει το θέμα των τιμών παρέμβασης. Όσον αφορά τις αθέμητες πρακτικές, στο εμπόριο, οι προτάσεις μας για την βελτίωση της θέσης των αγροτών στην τροφική αλυσίδα, δηλαδή αυτές συζητούνται ήδη στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και χαίρομαι που η έκθεση που ψηφίστηκε με 600 ψήφους στην Ολομέλειά σας αποτελεί και για μας σοβαρό κίνητρο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό και να το επιτύσσουμε στο μέλλον. Το θέμα της δίκαιης θέσης των αγροτών στην τροφική αλυσίδα για μας είναι, όπως είπα, από τα πιο σημαντικά θέματα. Στην αρχή τώρα της Σλοβακικής Προεδρίας διεξαγάγαμε διάσκεψη εμερογνωμόνων για το θέμα αυτό τα αποτελέσματα ή τα πορίσματα αυτής θα υποβληθούν στους υπουργούς στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Και θα συνδεθούν και με την αναμενόμενη έκθεση της Task Force. Στο τέλος της Προεδρίας μας ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε στο Συμβούλιο συμπεράσματα σχετικά με το θέμα αυτό. Ένας αριθμός από εσάς τους ευρωβουλευτές με ρωτήσατε σχετικά με συμφωνίες διεθνούς εμπορίου. Βεβαίως η Γεωργία παίζει σημαντικό ρόλο και μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εμπορίου. Σας διαβεβαιώ ότι το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο ε, σοβαρότατων συζητήσεων μεταξύ των Υπουργών Γεωργίας στο Συμβούλιο θα ανοιχθούν αγορές για την εξαγωγή προϊόντων. Αυτό είναι θετικό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγός αγροτικών προϊόντων στον κόσμο και υπάρχει δυναμικό και περαιτέρω ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, ή μάλλον οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων μπορούν να συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση τη κρίση στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ αλλά και με τι χώρε Μερκοσούρ θα αποτελέσουν αντικείμενο προσοχής από το Συμβούλιο και εμείς επιθυμούμε ε, να διασφαλίσουμε ότι θα είναι απολύτως ισορροπημένες οι διαπραγματεύσεις. Είναι ξεκάθαρη η εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει και τις προθεσμίες, αλλά και τις κόκκινες γραμμές που δεν επιτρέπεται να υπερβεί. Θα φροντίσουμε να μην μείνει ο μεγάλος χαμένος η αγροτική οικονομία των ε, συμφωνίων των συμφωνιών ελευθερίου εμπορίου. Και ιδίω για ευαίσθητα προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τι ΗΠΑ και το Μερκοσούρ, δηλαδή τι συμφωνίε με τι χώρε αυτέ, οφείλουμε να μην δυσμονούμε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ανταγωνιστικού εταίρου και έχουν και αυτοί επιθετικά εντό εισαγωγικών συμφέροντα, όπω και εμεί. Εμείς δεν θέλουμε η Γεωργία βεβαίως να θυσιαστεί για να κερδίσουμε πλονεκτήματα σε άλλους τομείς. Από την άποψη αυτή έγινε και μια ερώτηση για την σόρευση των διεθνών συμφωνιών. Οι σορευτικές επιπτώσεις, η σχετική μελέτη δηλαδή, θα δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο και ασφαλώς θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο ή του Συμβουλίου Υπουργών. Άλλο ενδιαφέρον θέμα που μου θέσατε και που απαντήθηκε ήδη μερικώς είναι η Βρετανική έξοδος. Προφανώς θα το συζητήσουμε αυτό, το Brexit. Πάντως εξ όσων γνωρίζω εξακολουθεί η Βρετανία να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσο παραμένει πλήρες μέλος έχει όλα τα δικαιώματα και φέρει όλε τι υποχρεώσει που συνεπάγεται η ιδιότητα μέλου και με τον τρόπο αυτό τι μεταχειριζόμαστε στο Συμβούλιο. Άλλη προτεραιότητα για μα είναι η δασοκομεία. Η κυρία Κέστινγκερ αλλά και άλλοι συναδελφοί σα έφυξαν το θέμα τη δασοκομεία. Χθε στην συνάντηση του προγεύματο μου είπαν ότι η δασοκομεία είναι ένα σημαντικό θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, έχει πρωτοπόρο ρόλο και για την αηφόρο ανάπτυξη της δασοκομείας. Και σε διεθνείς οργανισμούς θα προωθήσουμε την θέση αυτή, διότι η βιωσιμότητα της δασοκομείας έχει άμεσο ρόλο να παίξει στην προστασία του κλίματος. Στη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας θα διεξαχθούν δύο σημαντικές διεθνείς συναντήσεις για τα δάση, αφενός των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η Επιτροπή Δασοκομείας του ΦΑΟ. Εμείς θα καταλήξουμε σε κοινέ θέσεις με τις οποίες θα πάμε στις συναντήσεις αυτές. Ο ρόλος της Προεδρίας μας θα είναι ταυτόχρονα να επιμείνουμε στις θέσεις μας αυτές στις δύο προαναφερθείς συναντήσεις. Αναμένουμε και προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην δασοκομεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτάσεις, για παράδειγμα, για την ολοκλήρωση του Λουλουσιεφ στο γύρω στον ε, κύκλο προστασίας του κλίματος καθώς και τη χρήση δασοκομικών προϊόντων για παραγωγή ενέργειας. Θα προωθήσουμε λύσεις που να σέβονται τον πολυλειτουργικό ρόλο της δασοκομείας και της ε, βιώσιμης δασοκομείας. Γνωρίζουμε ότι συνεργάζεστε και με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασοκομείας. Θα διεξαγάγουμε και εμείς ειδική εκδήλωση για τη λειτουργία της δασοκομείας και του τομέα της ξυλίας. στα πλαίσια των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την Συμφωνία των Παρισίων. Αυτό θα γίνει τον Οκτώβριο και θα σας προσκαλέσουμε βεβαίω στην ε, διάσκεψη αυτή. Άλλο ενδιαφέρον θέμα που θέσατε είναι η κοινή αγροτική πολιτική και η απλούστευσή της. Απλούστευση της ΚΑΠ είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου εδώ και μια διετία. Και εμείς θα εγγύψουμε στο θέμα αυτό. Ωστόσο δεν είναι θέμα το οποίο ενδιαφέρει μόνο το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι θέμα το οποίο πρωτίστως ενδιαφέρει τους γεωργούς, τους αγρότες διότι η υπερβολική γραφειοκρατία δένει τα χέρια των αγροτών και η υπερβολική γραφειοκρατία και η γραφειοκρατική επιβάρυνση αυξάνει και το κόστος λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και οδηγεί και σε αστάθεια των τιμών των μεμονωμένων προϊόντων. Αμέσως μετά από την τελικοποίηση της δύσκολης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, τα συμμετέχοντα μέρη αντιλήφθησαν ότι το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη γεωργία περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία στη μεταρρύθμιση θεσπίστηκαν κανόνες με τρόπο που επιβάλλει ωστόσο βαριά γραφειοκρατικά άχθη στους αγρότες. Θα πρέπει τώρα να αξιολογήσουμε το νέο πλαίσιο Ενδεχομένω να είναι πρόημο να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση του πλαισίου. Ωστόσο, υποστηρίζουμε το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην αναθεώρηση των τμήματων εκείνης νομοθεσίας που προκαλούν τι χέρεις τους γεωργούς. Θα παρακολουθούμε την διαδικασία αυτή και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε οποιαδήποτε θετική προσπάθεια απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου. Αυτό αναφέρεται και στο λεγόμενο πρασίνισμα και μέτρα πρασινίσματος. Ένα χρόνο μετά από την αρχή της εφαρμογής του πρασινίσματος δεν μπορούμε ακόμα να πούμε ότι δεν είναι αποτελεσματικό το πρασίνισμα. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιε είναι οι πραγματικές επιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν να κρίνουμε ένα χρόνο μόλις μετά εάν είναι θετικέ οι επιπτώσει στην φύση. Για παράδειγμα, η διατήρηση βιοποικιλότητας όπου εκεί τα μέτρα του πρασινίσματος προσφέρουν σημαντική βοήθεια. Είναι μεγάλο το δυναμικό του greening εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά. Εξαρτάται πώς εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες μέλη. Μπορούμε να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών. Ωστόσο, υπάρχει χώρος για βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων πρασινίσματος. Όπως είπα προηγουμένως, θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε προσπάθεια απλοποίησης των μέτρων πρασινίσματος επίσης. Άλλο σημαντικό θέμα το οποίο αφορά τους αγρότες είναι η βιολογική γεωργία. Ο εισηγητής σας κύριος Χόισλινγκ υπέβαλε ερωτήσεις σχετικά με τη βιολογική γεωργία. Η Σλοβακική Προεδρία θα συνεχίσει στην πορεία που χάραξε η Ολλανδική Προεδρία και θα συνεχίσουμε την συνεργασία που έχουμε στον φάκελο αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι έχει επιδειχθεί πρόοδο και ασφαλώς θα επιζητήσουμε περαιτέρω πρόοδο στο φάκελο αυτό. Επί του παρόντος έχουμε αξιολογήσει στο τεχνικό επίπεδο το μεγαλύτερο μέρος της προτινόμενης νομοθεσίας. Γνωρίζουμε ότι πολιτικά το θέμα είναι ευαίσθητο. Η θέση πάντως του Συμβουλίου από πολλές απόψεις προσεγγίζουν τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι τεχνικό και επομένως τα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς ώστε να καταλήξουμε σε διατυπώσεις που όντω θα ωφελήσουν ολόκληρο τον τομέα. Μαζί με τις αντιπροσωπείες προχωρούμε σε μια ανάλυση σε βάθος όλων των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί ως τώρα για να ε, διευκρινίσουμε και ποια θα είναι τα μελλοντικά βήματα που πρέπει να λυθούν. Θα συνεχίσουμε την συνεργασία αυτή και στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε το έργο στον φάκελο αυτό. Έχουμε διεξαγάγει και σε φιλική ατμόσφαιρα ανεπίσημες ε, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων. Ελπίζω δε ότι η συνεργασία μας θα οδηγήσει σε θετικά συμπεράσματα. Ελπίζω ότι απήντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Εάν όχι, τουλάχιστον θεωρώ ότι μπόρεσα να απαντήσω σφαιρικά στις ανησυχίες σας, ανησυχίες των Ευρωβουλευτών και εκφράζω την ευχή να αποδώσουν καρπούς οι προσπάθειές μας και να διευκολυνθεί η ζωή των αγροτών. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας και ευχαριστούμε που μας δείξατε την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων της Σλοβακικής Προεδρίας που θα ασκήσει αυτό το εξάμεινο την Προεδρία του Συμβουλίου. Ε, θα διαπιστώσετε και από τη συζήτηση ότι σας στηρίζουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση και θεωρούμε ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, θα είναι δύσκολη η Προεδρία σας, αλλά πολύ συχνά οι δύσκολες Προεδρίες είναι οι ενδιαφέρουσες. Και δεν σας εύχομαι καλές διακοπές, γιατί ξέρω ότι και εσείς και το επιτελείο σας και οι συνεργάτες σας θα εργαστούν και στις θερινές διακοπές. Εν πάση περιπτώσει, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και θα ήθελα να πω ότι εδώ και αρκετό καιρό είχαμε πολύ καλές επαφές με τους συνεργάτες σας και ευελπιστώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η αγαστή συνεργασία. Ε, όπως σας είπα, η υπουργός θα παραδώσει τώρα συνέντευξη τύπου οπότε θα την απελευθερώσουμε και εμείς θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρης διάταξης. Ευχαριστώ.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 Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να ξανακαθίσουν στις θέσεις τους για να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Και κυρίως τα γαλλικά πηγαδάκια εκεί στο πίσω μέρος της αίθουσας παρακαλώ να διαλυθούν και να καθίσουν όλοι. Très bien. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας προτείνω να συνεχίσουμε με το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης που σχετίζεται με την παρουσίαση της μελέτης ε, του θεματικού τμήματος ε, για τα προγράμματα εφαρμογής της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της περίοδου 2015-2020. Είχαμε ε, ζητήσει τη μελέτη αυτή για τα προγράμματα αυτά η μελέτη αυτή εξετάζει τις επιλογές που πραγματοποίησαν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες προετοιμάζοντας τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την ε, εν λόγω περίοδο. Η μελέτη επίσης συγκρίνει τις επιλογές αυτές με τις επιλογές της προηγούμενης περίοδου 2007 με 2013 και έχει κάποια συμπεράσματα, κάποια στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το μέλλον της, αγροτικής, της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ευχηθώ να καλωσορίσω τους ε, δύο ομιλητές, την κυρία Τζάνε Ντουαέρ που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Gloucestershire στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον κύριο Φραντσέσκο Ματίνα που εργάζεται στο Συμβούλιο Γεωργικής Πολιτικής της Ιταλίας. Πριν τους δώσω το λόγο να πω ότι έχουν 20 ε, λεπτά να μοιραστούν μεταξύ τους, δεν είναι πολύ ο χρόνος αλλά για να μπορέσει να γίνει η συζήτηση υπό καλές συνθήκες 40 ε, λεπτά με το σύνολο των βουλευτών και ώστε να μπορέσετε να απαντήσετε μετά και αν θελήσει να μιλήσει και η Κομισιόν η κυρία η συγγνώμη, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ε, εκπροσωπείται από τον κύριο Λόγκου, δίνω το λόγο λοιπόν στην κυρία Ντουάιερ μπορείτε να ξεκινήσετε και καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την έκθεση αυτή. Πρόκειται για μια προκαταρκτική ουσιαστικά εξέταση των επιλογών των κρατών μελών και των περιφερειών των κρατών μελών ε, σε ό,τι αφορά τις νέες πολιτικές ανάπτυξη πέθρου που θα ισχύσουν μέχρι το 2020. Η δομή της παρουσίασης προβλέπει μια σύντομη εισαγωγή της προσέγγισης και του περιεχομένου και μετά εξέταση των πορισμάτων της μελέτης. Καταρχήν να δούμε πώς έχουν αλλάξει οι κανονισμοί και το πλαίσιο για να αντιληφθούμε καλύτερα ε, αυτά που βλέπουμε όσο αναλύουμε τα νέα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου και να κατανοήσουμε τις επιλογές των κρατών μελών και τα αίτια που οδήγησαν στις επιλογές αυτές. Ε, κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των σχεδίων για την νέα περίοδο προγραμματισμού και των ε, τρόπων και σχημάτων δαπανών της προηγούμενης ε, περίοδου προγραμματισμού και είδαμε πώς έχουν αλλάξει τα σχέδια σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και εξηγούμε και τους λόγους που κατά τη γνώμη μου διέπουν αυτές τις αλλαγές. Ποιος είναι ο στόχος καταρχήν της μελέτης. Ο στόχος της μελέτης ε, ε, δόθηκε ήδη από τη Γεωργία. Συγκριτική αξιολόγηση των επιλογών. Δίνουμε έμφαση στις επιλογές, όχι τόσο στα στοιχεία. Και προσπαθούμε να κατανοήσουμε γιατί τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειές τους ε, έδωσαν προτεραιότητα σε συγκεκριμένους στόχους και όχι σε άλλους. Και επίσης ε, ε, προσπαθήσαμε να δούμε αν αντιλήθηκαν κάποια συμπεράσματα και ε, βγήκαν διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες. Επίσης ε, εξετάσαμε ποια αιτία είναι σημαντικά και ποιες επιλογές θα είναι σημαντικές στην επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά την ολοκλήρωση αυτής της περίοδου προγραμματισμού. Η σχετική σύντηση θα ξεκινήσει ήδη από το 2018. Πρόκειται για μια ομαδική προσπάθεια με επικεφαλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά συνεργαστήκαμε με τον Δ. Ματίνο από την ΚΡΕΑ της Ιταλίας, το Ινστιτούτο Τιούνιγκεν της Γερμανίας, με πλούσια εμπειρία για την περιφερειακή προσέγγιση της Γερμανίας. Επίσης, ε, ε, συνεργαστήκαμε με την Ίνρα, στην Τιζόν της Γαλλίας, αλλά είχαμε και ε, συνεδριάσεις ε, στην ε, Μαδρίτη, στην Ισπανία, για παροχή συμβουλών. Επίσης εξετάσαμε τη Σύμφωνη Ιστερικής Σχέσης, που προσπάθησαν να διερευνήσουν την συνοχή μεταξύ των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των προγραμμάτων χρηματοδότησης και των άλλων ταμείων, της περιφερειακής ανάπτυξης, το κοινωνικό ταμείο, το Ταμείο Αλίας και το Ταμείο Συνοχής. Εξετάσαμε τα σχέδια δαπανών σε σχέση με την προηγούμενη και τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Εξετάσαμε τα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο και για τις 28 χώρες μέλη και επίσης ε, ε, εξετάσαμε λεπτομερώς ε, τα κράτη-μέλη που έχουν και πολλά περιφερειακά προγράμματα, ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα ευρωπαϊκά προγράμματα αντικατοπτριζόταν και στις περιφερειακές επιλογές των κρατών μελών. Επίσης αναζητήσαμε αξιόπιστες και ποιοτικέ πληροφορίες από εμπειρογνώμονες με τους οποίους είχαμε μακρά συνεργασία από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας τη γνώμη τους για τα βασικά αίτια των αλλαγών και το σκεπτικό των αλλαγών, καθώς και τις προτεραιότητες, τους στόχους και τις ανησυχίες που διέπουν τα νέα προγράμματα. Οπότε, αν εξετάσουμε το πολιτικό πλαίσιο, είναι οι κανονισμοί, οι εφαρμοστικοί κανονισμοί και η όλη στήριξη της νέας πολιτικής, διαπιστώνουμε ότι οι αλλαγές δεν είναι ρηξικέλευτες σε σχέση με τον παρελθόν, αλλά μια φυσική εξέλιξη της προηγούμενης κατάστασης. Επίσης ε, έγινε μια αλλαγή του τρόπου σκέψης, εντάσσεται η αγροτική ανάπτυξη σε ένα πιο συνεπές πλαίσιο με την εξέταση όλων των πηγών χρηματοδότησης, ώστε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν με συμπληρωματικό τρόπο τα διάφορα ταμεία και κονδύλια. Ε, και αυτή είναι μια έφαση που δίνεται στην τελευταία περίοδο προγραμματισμού. Επίσης, ε, περάσαμε από τους τρεις βασικούς άξονες των προηγούμενων ε, προγραμμάτων ανάπτυξη πέθρου σε ένα τέταρτο άξονα και του leader και μια πιο στοχευμένη προσέγγιση γύρω από έξι προτεραιότητες. Κάτι που δίνει το μήνυμα στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη περισσότερο τις ανάγκες και το πώς θα τηρηθούν ε, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προτεραιοτήτων. Επίσης, το πολιτικό πλαίσιο για το σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων ε, η οικονομική κρίση οδήγησε στην απόφαση περικοπής της χρηματοδότησης της κοινής πολιτικής. Στις διαπραγματεύσεις όμως για τη μεταρρύθμιση προβλέφθηκε αρκετή ελαστικότητα ώστε να μπορέσουν τα κρατημέλη να επιλέξουν ε, τον τρόπο αντίδρασης τους στην κρίση. Και έτσι ε, τα αρχικά κονδύλια για τα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου ήταν αρχικά χαμηλότερα από ό,τι στην προηγούμενη περίοδο, αλλά εξαιτία ή χάρη σε αυτή την ελαστικότητα και τη διακριτική ευχαίρεια ό,τι αφορά τη μεταφορά των κονδύλιων από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα, ε, σε σχέση με τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων και τις επιλογές χρηματοδότησης και εθνικής συμπληρωματικής χρηματοδότησης, τελικά το συνολικό αποτέλεσμα έδωσε στα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου στην τελευταία κρίση να είναι υψηλότερα για το σύνολο των 28 χωρών μελών σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Αν δούμε όμως την ισορροπία της χρηματοδότησης ε, μεταξύ των κρατών μελών επίσης έχει αλλάξει. Σε μερικές χώρες είχαμε μειώσεις και σε άλλες αυξήσεις της χρηματοδότησης. Και αυτό επηρέασε τις επιλογές των κρατών μελών για παράδειγμα, αν δούμε μια χώρα με αισθητέ περικοπές του προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε ότι η χώρα αυτή ε, προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο τον προγραμματισμό και υιοθετεί μια πιο στοχευμένη προσέγγιση. Ενώ χώρε που είχαν αύξηση κονδύλιων μπορούν να δείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία στους στόχους τους. Άλλωστε είναι αναμενόμενες αυτές οι συμπεριφορές. Σε ό,τι αφορά τα νέα στοιχεία του κανονισμού. Ο κανονισμός μοιάζει με το προηγούμενο, αλλά δίνει νέα έμφαση στη συνεργασία και στην προσπάθεια σχεδιασμού και εφαρμογής συνεργατικών προγραμμάτων και σχεδίων, ώστε να αυξηθεί ο αντικτυπός τους και η επίδρασή τους σε σχέση με το παρελθόν. Και επίσης ε, δίνεται ε, νέα έμφαση στην καινοτομία και στις εταιρικέ σχέσεις που ενισχύουν την καινοτομία. Ενθαρρύνονται οι γεωργοί να συνεργαστούν με ερευνητικά κέντρα ώστε να καινοτομήσουν ε, και να κάνουν πιο ανθεκτικό και βιώσιμο τον κλάδο τους στο μέλλον. Για παράδειγμα, το προηγούμενο μέτρο της πρόορης αξιοδότησης αφαιρέθηκε από το μένου των επιλογών και τα έκτακτα μέτρα που είχε η προηγούμενη περίοδος προγραμματισμού για να ε, διευκολύνει την ενταξιακή διαδικασία για τα κράτη-μέλη προσχώρησαν στην περίοδο 2004-2007 και αυτά τα μέτρα αφαιρέθηκαν γιατί ολοκληρώθηκε η ενταξιακή διαδικασία. Επίση είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι παρόλο που το πλαίσιο είναι πιο ελαστικό για τα κράτη-μέλη και για τον τρόπο που ανταποκρίνονται με στρατηγικό τρόπο στι ανάγκες και στις προτεραιότητές τους. Ο μηχανισμός με τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η ελαστικότητα έχει γίνει πιο περίπλοκος. Θα επανέλθω στο σημείο αυτό αργότερα γιατί επηρέασε αυτή η περιπλοκότητα, τις επιλογές των κρατών μελών. Ας δούμε τώρα τις αλλαγές στους πόρους. Βλέπετε από τη διαφάνεια τις δημοσιονομικές αλλαγές σε σχέση με την παλιά και τη νέα περίοδο προγραμματισμού για τη χρηματοδότηση των πυλών 1 και 2 της γεωργικής πολιτικής. Κάποια κράτη-μέλη αύξαν τους προϋπολογισμούς ανάπτυξης υπαίθρου, αλλά μείωσαν τους προϋπολογισμούς άμεσων ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα της πολιτικής. Και αυτό φυσικά επηρέασε τις επιλογές τους. Άλλες χώρες α, αύξησαν τα κονδύλια και στους δύο πυλώνες. Ενώ μερικέ αύξησαν τα κονδύλια είτε στον ένα κλάδο είτε στον άλλο. Είτε στην ανάπτυξη πέθρου είτε στις άμεσες ενισχύσει. Και άλλες χώρες μείωσαν τα κονδύλια και στι δύο πυλώνες. Όλα αυτά επηρέασαν τι επιλογές του φυσικά. Κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι οι δαπάνε δεν ήταν ε, ίδιε από την αρχή. Αν συγκρίνουμε για παράδειγμα τη σχετική ένταση πληρωμών και δαπανών ε, σε σχέση με την ε, επιφάνεια κάθε χώρας, την έκταση κάθε χώρας, βλέπετε από τους χάρτες ότι είναι διαφορετική ένταση των δαπανών. Μερικές φορές ε, αυτή η διαφορά οφείλεται σε ιστορικούς λόγους ή κάποια πολιτικά κριτήρια που επικρατούσαν κατά τη στιγμή της ένταξης σε σχέση με σήμερα, αλλά αυτή είναι μια διαδικασία που προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη, που προσπάθησε να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε αναθεώρηση των προγραμμάτων. Τώρα, για να δούμε τα νέα προγράμματα και τις προτεραιότητες. Οι έξι στρατηγικές προτεραιότητες που προσδιορίζονται, που καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προβλέπουν μόνο για πέντε ε, προτεραιότητες συγκεκριμένα κονδύλια. Η πρώτη προτεραιότητα που είναι η αλλαγή της γνώσης είναι μια προτεραιότητα που δρομολογείται μέσω των υπόλοιπων πέντε. Οπότε ε, η κατάρτιση, οι συμβουλές και η αφύπνιση είναι κάτι που επιδιώκεται μέσω των άλλων προτεραιοτήτων. Γι' αυτό και εξετάζουμε τις επιλογές των πέντε προτεραιοτήτων. Αυτός ο χάρτης δίνει και τον όγκο των πόρων στα κράτη-μέλη, αλλά και τις σχετικές ε, κατανομές κονδυλίων αναπροτεραιότητα. Ενδιαφέρον αυτό γιατί βλέπετε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ευρώπης ή των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Σκανδιναβικέ χώρες, δηλαδή στο Βορρά και στη Δύση, ιδιαίτερη έφαση στο περιβάλλον. Αυτή είναι η πρωταρχική προτεραιότητα των προγραμμάτων ανάπτυξη πέθρου. Ενώ σε χώρες όπως η Βουλγαρία ή η Ρουμανία, αλλά και στην Ανατολική και Βόρεια Γερμανία, δίνεται περισσότερη έμφαση στην ευρύτερη αγροτική ανάπτυξη και στην, ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην Ήπεθρο, τα θέματα του κοινωνικού αποκλεισμού και γενικώ κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονται. Άλλα κράτη δίνουν έμφαση στην ανταγωνιστικότητα στη Γεωργία, για παράδειγμα η Πολωνία ή κάποιες βαλτικές χώρες. Επίσης ε, αυτή είναι προτεραιότητα στην Πορτογαλία και σε κανένα δύο άλλες χώρες. Άλλες δύο προτεραιότητες ε, καταρχήν, η γεωργία που θα αντέχει στις κλιματικές αλλαγές. Η η τρίτη προτεραιότητα που αφορά τις τροφικές αλυσίδες και την διαχείριση του κινδύνου δεν χρησιμοποιούνται τόσο ευρέως στα κράτη-μέλη. Άντως, ο στόχος του κλίματος λαμβάνεται υπόψη κυρίως στις χώρες του Νότου και δικαίως στην Ισπανία, για παράδειγμα, την Πορτογαλία, τη Μάλτα. Εκεί μεγάλο τμήμα των μέτρων περιλαμβάνουν αυτή την περιβαλλοντική προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τη τροφική αλυσίδα και τη διαχείριση κινδύνου, αυτό είναι προτεραιότητα κυρίω τη Ιταλία. Είναι μια προτεραιότητα παλιά για του Ιταλού και ήταν ανέκαθεν σημαντικό αυτό ο τομέα. Τώρα, αν εξετάσουμε το περιφερειακό επίπεδο των χωρών που έχουν και πολλά περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξη πέθρου, ε, καταλήγουμε σε αυτό τον χάρτη που κατέρτισε το Ινστιτούτο Τιούνιγκεν της Γερμανίας και που ταξινομεί με διαφορετικό τρόπο τα μέτρα, όχι μόνο σε σχέση με τις στρατηγικές προτεραιότητες, αλλά και σε σχέση με τους ε, σκοπούς του σε περιφερειακό επίπεδο. Εκεί βλέπουμε άλλες διαφορές. Και κάποια νότια κρατήδια της Γερμανίας δίνουν έμφαση στο περιβάλλον, ενώ βόρεια και ανατολικά κρατήδια δίνουν περισσότερη έμφαση στην ευρύτερη ανάπτυξη της υπαίθρου. Ε, βλέπετε όμως κάποιο σχετισμό μεταξύ των προτεραιοτήτων και της οικονομικής κατάστασης των κρατηδίων. Γενικώ πάντως, εξετάζοντας την επιλογή των μέτρων των νέων προγραμμάτων, διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη επικεντρώνουν περισσότερους ε, πόρους σε μικρότερο αριθμό μέτρων σε σχέση με το παρελθόν. Επίσης, ε, βλέπουν ποια ήταν τα διδάγματα του παρελθόντος και επικεντρώνουν τους πόρους τους ε, σε λίγα σημαντικά σημεία. Και αυτό το γράφημα δείχνει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις 28 με, χώρες μέλη ε, τι ε, βάρος έχουν, οι κάθε, τι βάρος έχουν διάφορες προτεραιότητες. Και βλέπουμε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι το μέτρο που απορροφά περισσότερα κονδύλια. Επίσης, τα περιβαλλοντικά μέτρα ή τα μέτρα που έχουν περιβαλλοντικό στόχο ε, είναι σημαντικά. Η δεύτερη ε, προτεραιότητα σε ιεράρχηση, ε, δηλαδή μέτρα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Είναι τα δύο μέτρα αυτά τα πρώτα, τα περιβαλλοντικά και τις ανταγωνιστικότητες, απορροφούν τους μισούς πόρους του συνόλου των προγραμμάτων. Και φυσικά υπάρχουν, όπω σα είπα, διαφορέ μεταξύ των κρατών μέλων, όπω και στι στρατηγικέ προτεραιότητε. Τώρα βλέπουμε την αλλαγή στην κατανομή των κονδυλίων μεταξύ παλιά και νέα περίοδου. Τα τρία βασικά μέτρα αφορούν μεγάλε μεγάλες δαπάνες και στις δύο περιόδους. Το σύνολο, το άθροισμα έχει μειωθεί, αλλά αυτό αφορά και την περίοδο προγραμματισμού του προϋπολογισμού. Πάντως υπάρχει αισθητή μείωση στις επενδύσεις στα δάση ε, σημαντική μείωση σε κάποια μέτρα ευρύτερης αγροτικής ανάπτυξης προηγούμενης περίοδου, ε, ενώ αντίθετα έχουμε αισθητή αύξηση των κονδυλίων του Λίντερ. Και αυτό γιατί ο νέος κανονισμός απαιτεί από τα κράτη-μέλη να δαπανίσουν 5% των κονδυλίων στο Λίντερ. Ενώ στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού η απέτηση ήταν 3%. Ενώ για τα παλιά κράτη ήταν 5% και για τις δύο περίοδους. Τα άλλα νέα μέτρα, διαχείριση του κινδύνου, το, σχετικό κονδύλιο αυξήθηκε γιατί αρχικά ήταν στον πρώτο πυλώνα της πολιτικής και το, άρθρο το μέτρο 16 της συνεργασίας με πολλές επιλογές προωθείται κυρίως στο νέο πλαίσιο και εφαρμόζεται με πολύ θετικό τρόπο. Εξετάσαμε τις αλλαγές μεταξύ των δύο περιόδων και εξετάζοντας την έκταση στην οποία αλλάζει σημαντικά το επίπεδο του κράτους μέλους ή αν ο κόσμος παραμένει σε αυτά που γνωρίζει. Στον πίνακα αυτό γίνεται μια προσπάθεια να δείξουμε με σύντομο τρόπο τομείς ε, όπου υπάρχει συνοχή ή αλλαγή μεταξύ των δύο περίοδων. Οπότε τα ροζ τετράγωνα εδώ δείχνουν τις χώρες που δεν άλλαξαν πολύ τις στρατηγικές τους όσον αφορά την κατανομή των πόρων μεταξύ περίοδων στα πράσινα πλαίσια Βλέπουμε χώρες που έκαναν μια αλλαγή προς ε, περισσότερο περιβαλλοντικούς σκοπούς και τα πορτοκαλί πλαίσια είναι τα λίγα κρατημέλη όπου βλέπουμε να κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση λιγότερο περιβαλλοντικά και είτε ευρύτερη η αγροτική ανάπτυξη είτε ανταγωνιστικότητα. Και όπως βλέπετε είναι μια συντηρητική εικόνα γενικά, αλλά υπάρχουν και ενδιαφέρουσες κινήσεις. Ε, λίγο περισσότερη εστίαση στο περιβάλλον από ό,τι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Το ίδιο κάναμε και σε περιφερειακό επίπεδο στις χώρες όπου υπάρχουν πολλά περιφερειακά προγράμματα. Και εδώ έχουμε ένα παρόμοιο πίνακα για τις περιφερειές της Ιταλίας, όπου βλέπουμε πολλές που βρισκόνται στη μέση, στα ροζ πλαίσια που δεν άλλαξαν ιδιαίτερα, αλλά κάποιες άλλαξαν όσον αφορά τις προτεραιότητες που έθεσαν. Και πάλι πολλές ε, περιφέρειες έδωσαν μεγαλύτερη προτεραιότητα στο περιβάλλον από ό,τι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Κοιτώντα τα περιφερειακά RDP, τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, ε, έγινε ανάλυση σε τέσσερα κράτη-μέλη και τα μοτίβα μοιάζουν με αυτά που βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά αντιλαμβανόμαστε λεπτομερώς και τις αιτίε, γιατί έχουμε εμπειρογνώμονες στα κράτη-μέλη αυτά. Έγινε μια συζήτηση για το ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν σε τέτοιες αλλαγές. Παρατηρούμε το στην Ιταλία στη Γερμανία, ότι εκεί όπου οι περιφέρειες ε, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες οικονομικής ανάπτυξης και μείωση της ενεργείας, η στρατηγική αφορά ευρύτερη επένδυση στην αγροτική οικονομία. Ενώ στην Ισπανία γίνεται συνειδητά η επιλογή ότι οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα ε, αντιμετωπίζονται με σημαντικές γεωργικές επενδύσεις, δηλαδή διαφορετικός τρόπος απόκρισης ε, για την κάλυψη των αναγκών στις διάφορες χώρες. Επίσης παρατηρούμε και κάποιες αποκρίσεις όσον αφορά το συνδυασμό ε, της πολυπλοκότητας των διαφόρων κανονισμών. Στις πιο εύπορες περιοχές ε, υπάρχει αίσθηση ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα με πιο περίπλοκο ή πιο δύσκολο τρόπο. Στη Γερμανία, το, οι εμπειρογνωμόνες του Ιδρύματος Turing μας εξήγησαν ότι κάποια από τα μέτρα δεν προγραμματίζονται πλέον στο πλαίσιο των προγραμμάτων ε, αγροτικής αναπτύξης, απλά λαμβάνονται υπόψη ως ε, κρατικές ενισχύσεις ε, στις χώρες αυτές, γιατί θεώρησαν οι αρχές ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ορισμένα δύσκολα πράγματα μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου, γιατί είναι πολύ επαχθές. Πολύ δύσκολο στην εφαρμογή. Οπότε τρέχουν ως εθνικά προγράμματα. Αυτό πιστεύω είναι σημαντικό να το παρατηρήσουμε. Στη Γαλλία από την άλλη, όπου υπάρχουν περισσότεροι πόροι, υπάρχει και μεγαλύτερη δέσμευση χρήση αυτών των πόρων στα προγράμματα ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά χρηματοδότηση και να γίνουν περισσότερα. Στην Ιταλία, με πολύ ενδιαφέρον παρατηρούμε ότι κάποιες βόρειες περιοχές της Ιταλίας καινοτομούν Μίλησε για τις στρατηγικές προτεραιότητες ε, της Ιταλίας ε, για τα μέτρα ε, της τροφικής αλυσίδας και τη χρήση των νέων μέτρων συνεργασίας. Θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι καινοτόμα και πολύ ενδιαφέροντα. Προσπαθήσαμε να, με μια απλή άσκηση να εξετάσουμε την έκταση στην οποία συγκρίνοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πόροι φαίνεται να ακολουθούν ή όχι τις σχετικές ανάγκες. Είναι μια απλή άσκηση και σίγουρα απλουστεύει πολύ το τι θα θεωρήσουμε ως δείκτες ανάγκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ισχυρότερη σχέση που βρήκαμε μεταξύ προτεραιοτήτων κράτους μέλους και δικτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για σχετικές ανάγκες ήταν η εξής. Αφορά τους ανθρώπους σε κίνδυνο φτώχεια ή κοινωνικού αποκλεισμού σε αγροτικές περιοχές που είναι ένα σύνολο δεδομένων που έχει ε, συγκεντρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό το συγκρίναμε με το βαθμό στον οποίο τα προγράμματα έδωσαν προτεραιότητα στην ευρύτερη αγροτική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη. Και υπάρχει μια θετική έσκηση, διαφάνεται πιθανώ εκεί, όπου οι χώρε με τι μεγαλύτερε ανάγκε προγραμμάτισαν πιο ισχυρά αυτή την προτεραιότητα. Αλλά κοιτώντα άλλε προτεραιότητε είναι πιο δύσκολο να δείξουμε τη σχέση ή να αποδείξουμε ότι η σχέση είναι σωστά θεμελιωμένη. Υπάρχουν και πολλοί, ε, στο, πολλοί, πολλοί λόγοι που αφορούν τις συνθήκες, τις τοπικές συνθήκες. Ε, αλλά βλέπουμε εδώ τη σχετική, τη σχετική σπουδαιότητα περιβαλλοντικά ορισμένων περιοχών και τις προτεραιότητες που επιλέγησαν. Ε, πώς χρηματοδότηση δόθηκε σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Ε, όσο πιο προστατευμένη μια περιοχή φαίνεται, τόσο λιγότερα χρήματα δίνονται για το περιβάλλον. Ίσως να έχει μια λογική αυτό βέβαια. Μετά κοιτάξαμε τη σχέση μεταξύ της ε, ανταγωνιστικότητας ως προτεραιότητας ε, και των μέτρων σχετικής ε, ανταγωνιστικότητας ευρωπαϊκό επίπεδο και εκεί δεν βρήκαμε καμία σχέση. Όπως φαίνεται άλλα πράγματα αιτιολογούν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση προς την γεωργική ανταγωνιστικότητα από οποιαδήποτε επισκόπηση των σχετικών αναγκών. κάποια επιχειρήματα δυνατοτήτων ίσως να είναι πιο ισχυρά από τα επιχειρήματα των αναγκών στο πλαίσιο αυτό. Τώρα κάποια συμπεράσματα. Σας ενθαρρύνω αν προλάβετε να διαβάσετε τα συμπεράσματα της έκθεσης τα οποία πάνε σε μεγαλύτερο βάθος και να δείτε και κάποια από τα σκεπτικά που παρουσιάζουμε πιο λεπτομερώς. Συνολικά, η αποκρίση στο νέο πλαίσιο, στο νέο κανονισμό και στη νέα προγραμματική περίοδο υπήρξε αρκετά συντηρητική. Πολλά κράτη-μέλη δηλαδή φαίνεται να λένε κρατάμε τα πράγματα όπως έχουν. Κάνουμε αυτά που, έχουμε γνωρί, που γνωρίζουμε ήδη. Αν δείτε το μοτίβο των δαπανών σε μέτρα, σε κάποια μέτρα, είναι περισσότερα τα μέτρα στα οποία μειώθηκαν οι δαπάνες, οπότε υπάρχει κάποια απαγίωση στο να μπαίνουν λιγότερα χρήματα σε λιγότερα μέτρα, περισσότερα προγράμματα. Και επίση φαίνεται να υπάρχει απομάκρυνση από τη χρήση τη χρηματοδότηση τη κοινή γεωργική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη. Σε κάποια νέα προγράμματα πραγματικά τελικά το Leader είναι το μόνο εργαλείο το οποίο προωθεί την ευρύτερη αγροτική ανάπτυξη πέραν των ε, άλλων πόρων οι οποίοι ε, δρομολογούνται προς την ε, διαχείριση του περιβαλλοντος και το γεωργικό τομέα. Ο νέος κανονισμός της Κομισιόν προσέφερε πολλά νέα εργαλεία ανέφερα τη διαχείριση κινδύνων. Υπήρχε και η δυνατότητα να τρέξει κανείς υπό προγράμματα για συγκεκριμένους τομείς ε, με πολύ εξειδικευμένες προσεγγίσεις. Υπήρχε, η δυνατότητα χρήσης ε, χρηματοδοτικών μέσων για πρώτη φορά. Μεταξύ όλων αυτών των επιλογών, όπως φαίνεται, ελάχιστες ε, έγιναν δημοφιλείς μεταξύ των διαχειριστικών αρχών που σχεδιάζουν τα προγράμματα. Το μέτρο συνεργασίας αποτελεί εξαίρεση διότι οθετηθήκε σε μεγάλο βαθμό, χρησιμοποιήθηκε με πάρα πολλού τρόπου σε πολλά κράτη-μέλη και κάνουμε μια ανάλυση για αυτό το μέτρο στην έκθεσή μα. Αλλά η διαχείριση κινδύνων δεν χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα. Τα θεματικά υποπρογράμματα πιστεύω δεν επιλέγησαν διότι θεωρήθηκαν ω άλλη μια στρώση γραφειοκρατία ε, στον ήδη πολύπλοκο προγραμματισμό και τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα. Όταν ρωτήσαμε τι επαφέ μα στα κράτη-μέλη για τι κυρίε επιρροέ και ε, τους κινητήριους μηχανισμούς φαίνεται ότι αποκομίστηκαν κάποια διδάγματα από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους τι λειτουργεί καλά, τι μπορούμε να διαχειριστούμε εύκολα, τι είναι περίπλοκο και σίγουρα υπήρξε και η επιρροή της οικονομικής κρίσης όπως είπε και ένας από τους προηγούμενους ομιλητές τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί, που μπορεί ή όχι να σχετίζονται με την κλιματική αναλογή ε, οδηγούν σε διαφορέ όσον αφορά τον ορισμό προτεραιοτήτων για το μέλλον. Επίση, ακούσαμε ότι η Κομισιόν επηρέασε σημαντικά τα προγράμματα, ειδικότερα στο να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη και ε, ότι ενσωματώνουν κάποια ε, την περιβαλλοντική διάσταση και ορισμένα συγκεκριμένα λόμπι σε ορισμένε ε, χώρε επισημάνθηκαν ω λόμπι που επηρεάζουν ιδιαίτερα τη διαδικασία. έχουμε περισσότερα στοιχεία συντονισμού της χρηματοδότησης μεταξύ των, ε, της αγροτικής ανάπτυξης ε, μέσω της, ε, των γεωργικών ταμείων και των άλλων ταμείων και είχαμε και κάποια για το σχεδιασμό στις συγκεκριμένες περιοχές και είχαμε και το μέτρο 16 για τη συνεργασία, αλλά δεν μπορούμε τώρα να βγάζουμε συμπεράσματα για την καινοτομία. Σε δύο-τρία χρόνια θα δούμε κατά πόσο αυτές οι νέες επιλογές οδήγησαν σε καινοτομία ρεαλιστική. Αλλά πιστεύω ότι και η δουλειά που έχει γίνει στη διατροφική αλυσίδα είναι ενδιαφέρουσα. Καλό θα να δούμε τι έκαναν οι Ιταλικές περιφέρειες σε αυτό το θέμα. Συνολικά, ωστόσο, πιστεύω, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι η Κομισιόν προσπάθησε μέσω αυτού του κανονισμού να δημιουργήσει κάτι πιο ευέλικτο, πιο προσαρμόσιμο στις τοπικές συνθήκες και που θα επέτρεπε πιο στρατηγική και αποτελεσματική ως προς το κόστος χρήση των πόρων, αλλά ταυτόχρονα έφτιαξαν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο πλαίσιο, τόσο για την προετοιμασία των προγραμμάτων, όσο και για την επακολούθη εφαρμογή, παρακολούθηση και για την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων. Και αυτό που με ανησυχεί ότι είναι ότι αν αυτό αρχίσει να επηρεάζει το σχεδιασμό και τη λειτουργία των προγραμμάτων, θα αποτελέσει εμπόδιο για την επίτευξη πραγματικής πρόοδου μας αυτών των ταμείων. Αν λοιπόν οι διαχειριστικές αρχές ε, ε, αρχίσουν να ε, ρίχνουν χρήματα σε τομείς όπου οι δαπάνες είναι εύκολες αντί για τις, τους τομείς όπου χρειάζονται περισσότερο τα πράγματα είναι ανησυχητικά ε, κάποιες χώρες έχουν λάβει μικρότερο προϋπολογισμό για τις άμεσες ενισχύσεις και εκεί υπάρχει μια τάση χρήσης ε, της χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη ως αντιστάθμισμα για αυτή, το μικρότερο ποσά. αν τώρα η Επιτροπή αναρωτιέται ποια θα πρέπει να είναι νέα μεταρρύθμιση, νέε μεταρρυθμίσει, πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση τη απλούστευση στο πλαίσιο τη πολιτική εστιάστηκε ιδιαίτερα στο πυλώνα 1 και στη διαταξία των greening. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να μα απασχολήσει και η αγροτική ανάπτυξη, η ανάπτυξη τη υπαίθρου. Αν δεν απλουστεύσουμε το πλαίσιο και δεν το διευκολύνουμε, δεν διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη να εκπληρώσουν τι φιλοδοξίε του και να δείξουν δημιουργικότητα για να καλύψουν τι τοπικέ και περιφερειακέ ανάγκε, τότε δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις φιλοδοξίες της Ευρώπης για την αηφόρα ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική. Ευχαριστώ. Merci, merci à vous pour cette... ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την θαυμάσια αυτή παρουσίαση της εκθέσεως. Θα αρχίσουμε την συζήτηση. Η κυρία Πετήρ έχει ζητήσει να, να, μπορέσει να λάβει το λόγο για την έκθεση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, ε, να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες που έχουν ε, προβεί σε δελεχή ανάλυση των προγραμμάτων. Ξέρουμε ότι η Κροατία είναι νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι στιγμής δεν έχει απορροφεί σχεδόν κανένα κονδύλιο από τα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου και μάλιστα είχαμε και πρόβλημα γιατί ο πρώην υπουργό Γεωργίας προκήρυξε κανονισμό με το το σχήμα ουσιαστικά ουσιαστικά ευνόησε κάποιες ε, επιχειρήσεις ε, των συγγενών του και δεν έκανε ε, καλή κατανομή των κονδύλιων. Άλλαξε η κυβέρνηση, αλλά ο νέος υπουργός δεν ακύρωσε τον προηγούμενο διαγωνισμό και περίπου 500 εκατομμύρια ακούνα έχουν μείνει μπλοκαρισμένα, δεν έχουν φτάσει στους γεωργούς για την ανάπτυξη πέθρου και ταυτόχρονα δεν ξέρουμε πώς να λύσουμε την κρίση. Ποια είναι η δική σας συμβουλή. Από τη στιγμή που στην πρώτη προκήρυξη διαγωνισμού ε, υπήρξαν ατασταλίες, δεν πρέπει να ακυρωθεί ή να κάνουμε αυτό που επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκλειστούν οι επιχειρήσεις ε, που η συμμετοχή τους δεν ήταν σωστή ή προτείνεται κάποια τρίτη λύση. Πώς θα μπορούσαμε να εκταμιεύσουμε αυτά τα κονδύλια, να τα απεμπλέξουμε τη χρήση τους ώστε να μην τα χάσουμε τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, μας δείχνει πώς θα γίνει η κατανομή του χρόνου στην Ευρώπη και τι μπορούν να αναμένουν οι χώρες μέλη από τα προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ερώτηση. Κύριο θέμα τον τελευταίο αυτό καιρό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η κατάσταση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και όσον αφορά αθέμητες πρακτικές ανταγωνισμού. Από την άλλη μεριά υπάρχει το πρόβλημα της διαχείρισης των κινδύνων από την ε, σκοπιά των αγορών και βέβαια πάντοτε η αλλαγή του κλίματος. Κατά τη γνώμη σας, το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται επαρκώς στα προγράμματα ανάπτυξη της υπαίθρου. Γνωρίζω ότι εδώ ο πρώτος πυλώνας είναι σημαντικός. Είπατε ότι ιδίω για τις βόρειες ιταλικές περιοχές, οι περιφέρειες, είναι σημαντικό να εξεταστεί με ποιο τρόπο έχουν οργανωθεί. Διότι τα όσα συμβαίνουν στην αγορά και πώς οργανώνονται οι αγρότες και πώς οργανώνουν τις τροφικές αλυσίδες Αυτά είναι σημαντικά διότι εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα απέναντι στις αλλαγές. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να τονιστεί περισσότερο η ανάγκη ενίσχυσης της τροφικής αλυσίδας μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της υπαίθρου. Ευχαριστώ κύριε Μπόγκοβιτς. Ακόμη πέντε συναδέλφους έχω εγγεγραμμένους. όπως είπα πέντε, έχω πέντε πρόσωπα έχω και γραμμένα. Δεν θα σας περιορίσω το χρόνο, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομοι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη ζήτηση αυτή μέχρι τις 11.30. Κύριε Άγνιου. Μικρόφωνο. Εγώ δεν είχα ε, πρόθεση να μιλήσω, αλλά πάντως θα πάρω το λόγο. Δύο ερωτήσεις. Και οι δύο ερωτήσεις σχετικά με το κλίμα. Μήπως μπορείτε να επεκταθείτε με λίγες φράσεις και να με βοηθήσετε. Το πρώτο που είπατε ήταν ε, αγροτική οικονομία, η γεωργία, που να είναι ανθεκτική στις αλλαγές του κλίματος. Τι είναι αυτό και ε, τι χρήματα επενδύονται για να γίνει αυτό. Ε, πώς θα πρέπει εγώ να αλλάξω τα όσα κάνω στη γεωργική εκμετάλλευση ώστε να γίνει αυτή η ανθεκτική στις αλλαγές του κλίματος. Σε άλλη φράση χρησιμοποίησατε τη λέξη ενισχύσεις για το κλίμα, για τη Γεωργία. Τι ακριβώς είναι αυτές. Merci, Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντεκάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. βαθύνει σε πολλού τομεί με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Μία πολύ συγκεκριμένη τώρα ερώτηση. Ένα από τα θέματα που θίξατε είναι αυτή η συγκέντρωση των μέτρων, δηλαδή λίγα και σημαντικά μέτρα εντό των κρατών μελών. Αν αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε από τα μέτρα που ουσιαστικά υπαγορεύουν τα ευρωπαϊκά κριτήρια, δεν θα ήταν απλούστερο τα προγράμματα, οι χώρες που έχουν πολλά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ε, ε, τα κράτη-μέλη λεφτά να επικεντρωθούν σε εθνικά μέτρα τελικά στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών μέτρων σε όλες τις περιφέρειες, σε όλα τα λέντρα, τα κρατήδια της Γερμανίας. Δεν θα ήταν πιο απλό λοιπόν ε, ουσιαστικά να υπάρχει ένα ενιαίο μέτρο για όλες τις χώρες αντί να τα κατακαιρματίζουμε τα μέτρα μεταξύ περιφερειών αφού είναι περίπου τα ίδια. Ευχαριστούμε. Το, λόγο έχει ο κ. <clears throat> Ευχαριστώ για την παρουσίαση της ε, εκθέσεως. Βρήκα ε, ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες μέλη. Εγώ είχα κατανοήσει ότι ο δεύτερος πυλώνας λαμβάνει μάλλον μεγαλύτερη προτεραιότητα σε όλες τις χώρες μέλη. Διαπιστώνω τώρα από την μελέτη σας ότι έχει χάσει πολύ σε όγκο και δεν βρισκόμαστε λοιπόν πάνω σε ενιαία γραμμή. Είναι πολύ διαφορετικές οι προτεγγίσεις των χωρών μελών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση στην Ευρώπη. Το θετικό που μπορώ να πω είναι ότι τα μέτρα για την αγροτική οικονομία αυξάνονται, αλλά ίσως και εκεί μπορείτε να εξηγήσετε, διότι και εκεί υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Και τι ακριβώς σημαίνουν τα μέτρα αυτά. Είναι μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, είναι μέτρα προώθησης της βιολογικής γεωργίας, τα έχετε βάλει μαζί αυτά ή μήπως μπορείτε να κάνετε κάποια διαφοροποίηση. Και επίσης ε, τα κονδύλια για τα προγράμματα leader. Τι ρόλο παίζουν αυτά και θεωρείτε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο, θα πρέπει να, το οποίο η χρήση θα πρέπει να επεκταθεί. Και τέλος, οι προσπάθειες για τη δημιουργία κοινοπραξιών στις διάφορες περιφέρειες, για παράδειγμα πρωτοβουλίες για την διάθεση στην αγορά προϊόντων. Μπορείτε να πείτε ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε άλλες χώρες. Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη μελέτη. Πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτή η συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο θεμελιώδη ζητήματα και να ρωτήσω πώς επηρέασαν τα εθνικά αλλά και τα περιφερειακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Ε, είχαμε σημαντικές ενισχύσεις για την ένταξη των νέων στη Γεωργία. Πώς επηρέασαν ε, τα προγράμματα και τι έγινε με τη συγκέντρωση της προσφοράς. Γιατί και η στήριξη των νέων και η συγκέντρωση προσφοράς είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα και σημαντικές μας προκλήσεις. Πώς επηρέασαν συγκεκριμένα αυτά τα δύο θέματα τα προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριος Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Χόγκαν μιλάει συχνά για απλούστευση και στο δικό του κατάλογο προτεραιοτήτων προηγείται ο πρώτος πυλώνας. Κάτι που με ενοχλεί, γιατί εμείς προτιμούμε το πυλώνα 2, αν και πρέπει κανείς να έχει την ευφία και το δίκτυο νομοσύνης του Αϊνστάιν ή σχέση με τον Αϊνστάιν για να καταλάβει τα μέτρα γιατί είναι τόσο περίπλοκα. Πρώτα αυτό θα πρέπει να αναλύσουμε. Πού έγινε η περιπλοκότητα πριν προσπαθήσουμε να τα απλουστεύσουμε. Αλλά πραγματικά δεν έχω μέτρο σύγκρισης για να σας αποδείξω πόσο πραγματικά περίπλοκα είναι αυτά τα μέτρα. Ευχαριστούμε κύριε Φλάνναγκαν. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δώσω το λόγο και στους εμπειρογνώμονές μας, θα ήθελα και εγώ να κάνω λίγα σχόλια. Καταρχήν να σα ευχαριστήσω για την πολύ αξιόλογη μελέτη σας. Και να σας ρωτήσω, τι γίνεται με την ε, πολυταμιακή προσέγγιση, ελήφθη υπόψη στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ο συνδυασμός δηλαδή των διαφορών ταμείων. Επίσης, διαπιστώσαμε κάποια πρόοδο στις διάφορες, ε, στους διάφορους πίνακες ό,τι αφορά τη προσέγγιση. Δεν θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τέτοιου είδους ε, ολιστικές προσεγγίσεις και συνδυασμό των διαφόρων ταμείων. Και Στη μελέτη που κάνατε, δεν θα προτείνατε καλύτερη επανισορρόπηση μεταξύ των δύο πυλώνων, του πρώτου και του δεύτερου. Γιατί μερικές ε, επιλογές έμειναν ατελέσφορες ε, και του πρώτου πυλώνα που αφορά αμυγός ε, τη γεωργία και του δεύτερου που, αφορούν, που αφορά την αγροτική ανάπτυξη, την ανάπτυξη πέθρου. Αυτή θα είναι η ερώτησή μου και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λόγκο, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, σε περίπτωση που θέλει να σχολιάσει την ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω το ενδιαφέρον που έχουμε εμεί για αυτή τη ε, μελέτη που έγινε με τόση επιμέλεια. Θεωρούμε ότι είναι υψηλή ποιότητα ε, δουλειά που συμπληρώνει άρεστα τη δική μας εξάντε αξιολόγηση. Το δεύτερο που ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι επισημαίνεται ένα μέγιστο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία Λίντερ όσον αφορά τις ε, χρηματοδοτήσεις αλλά και για το μέτρο που αφορά τη συνεργασία δηλαδή για ολόκληρη την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί και η καινοτομία επίσης μας φαίνεται ένα θετικό σημείο. Το τρίτο θετικό σημείο της έκθεσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του προγραμματισμού από απόψη γενικής συνοχής των προγραμμάτων. Προφανώς ε, ε, αυτή η προσπάθεια είναι κάτι για το οποίο πρέπει να επενέσουμε τη κρατημέλη και τις περιφέρειες. Τέλος, ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο που χαρακτηρίστηκε ως αρνητικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα πλήρης χρήση των ε, χρηματοδοτικών μέσων. Εμείς θέλουμε να επιθυμίσουμε ότι έχουμε συνεργαστεί εντατικά με την ομάδα Bay την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να δημιουργήσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα και συνεργαζόμαστε με πολλές περιφερειές στην Ιταλία προσπαθώντας να αναπτύξουμε ένα εργαλείο ε, πολυπεριφερειακού χαρακτήρα που να μπορεί να παρέχει συνθήκες πρόσβασης σε πιστώσεις πολύ καλύτερες. Όσον αφορά την απλούστευση του δεύτερου πυλώνα, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του Επιτρόπου μου. Εμείς εργαζόμαστε εντατικά για συγκεκριμένες προτάσεις απλούστευσης. Και έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες, κύριε Πρόεδρε, προσπαθώντας να προσανατολίσουμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες προς μια απλούστερη υλοποίηση με πιο διαφανή, πιο απλά μέτρα, πιο ουσιαστικά μέτρα, τα οποία θα διευκολύνουν πρώτα απ' όλα τη ζωή των τελικών δικαιούχων. Και υπό αυτή την έννοια θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με μεγάλη δέσμευση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Euh, Ευχαριστώ αγαπητέ εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημαντικό είναι να εργαστούμε και ε, πάνω στα λογιστικά σχέδια των χώρων μελών. Να διευκολύνουμε επομένω την μελέτη της ερώτησης αυτή, του θέματος αυτού. Και την διαχείριση στο περιφερειακό επίπεδο των προγραμμάτων. Για να απαντήσετε σε, αυτή, ε, σε αυτό το πλήθος ερωτήσεων, ε, λαμβάνει το λόγο κυρία Ντουάιλερ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας. Επιτρέψτε μου να παρακαλέσω τον συνάδελφό μου Μαντίνο να απαντήσει σχετικά με την τροφική αλυσίδα για την Ιταλία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως υπόθηκε στην παρουσίαση της μελέτης, ένα από τα σημεία κλειδιά υπήρξε η προσοχή στη διατροφική αλυσίδα. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα στην Ιταλία, διότι στην Ιταλία έχουμε την παράδοση σχεδιασμού των παρεμβάσεων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης στις ε, αγροδιατροφικές αλυσίδες. Το εργαλείο αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον διότι μπορεί επίσης ε, να αποκριθεί σε ορισμένα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν σήμερα το πρωί κατά τη συζήτηση για την ε, εκ νέου εξισορρόπηση της κατανομής της αξίας εντός της αγροδιατροφικής αλυσίδας, διότι ποια είναι η καινοτομία που προσφέρουν αυτά τα προγράμματα, η καινοτομία τους της, στο πλαίσιο της αγροδιατροφικής αλυσίδας είναι ότι βρίσκουν ε, σημεία συμφωνίας μεταξύ της ε, πρωτεογενούς παραγωγής ε, και της αγροδιατροφικής βιομηχανίας όσον αφορά την ανάπτυξη των αλυσίδων. Και φυσικά και όσον αφορά και την οργάνωση των αλυσίδων, διότι η οργάνωση των αλυσίδων είναι ένα από τα δύναμα σημεία της ε, γεωργίας σε πολλές περιφέρειες. Αυτή λοιπόν η πτυχή Αποδείχθηκε ότι ήταν μια από τις σημαντικότερες πτυχές τόσο στην παλιά προγραμματική περίοδο και δεδομένη της επιτυχίας εκείνων των προγραμμάτων και στη μελλοντική, ε, στο μελλοντικό, στη μελλοντική προγραμματική περίοδο. Ήθελα να πω και κάτι όσον αφορά την απλούστευση. Μας ρώτησαν γιατί απλουστεύουμε το δεύτερο πυλώνα. Γιατί θα έπρεπε να τον απλουστεύσουμε το δεύτερο πυλώνα, ο οποίος είναι πιο απλός. Ουσιαστικά τρία είναι τα σημεία τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν όταν μιλάμε για απλούστευση. Συχνά λέμε ναι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη απλούστευση, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα γενικό σχόλιο αυτό. Πρέπει να εστιαστούμε λοιπόν σε τρία ζητήματα. Το πρώτο που ε, χρήζει απλούστευσης είναι οι σχέσεις μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα και ουσιαστικά μεταξύ greening και αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Διότι η Κομισιόν μας ζητά να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δύο και αυτός ο διαχωρισμός συνεπάγεται μια σειρά κανόνων και ελέγχων πολύ αυστηρών που τελικά περιπλέκουν εξαιρετικά το όλο ζήτημα. Όταν μιλάμε λοιπόν για απλούστευση το πρώτο πράγμα στο οποίο πρέπει να εστιαστούμε ε, είναι το ζήτημα της σχέσης μεταξύ του greening και των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Αν εμείς καταφέρουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, θα έχουμε κάνει μια μεγάλη χάρη προς τους γεωργούς. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που αφορά την απλούστευση είναι η σχέση μεταξύ πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και των πολιτικών συνοχής. Διότι ναι, μεν αυτές οι δύο πολιτικέ αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων, ωστόσο οι κανόνες μεταξύ του είναι εντελώ διαφορετικοί. Έχει σημειωθεί σίγουρα κάποια πρόοδο στη μεταρρύθμιση του 2007-2013, αλλά η πρόοδο αυτή δεν είναι επαρκής. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι ώστε οι κανόνε λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να είναι όσο το δυνατόν πιο όμοιοι. Γι' αυτό το λόγο η προσέγγιση πολλών ταμείων του Λίντερ δεν υιοθετήθηκε σε πολλές περιφέρειες, σε πολλές περιπτώσεις, διότι το να πρέπει κανεί να εργαστεί με τρία ταμεία που λειτουργούν το καθένα με διαφορετικό τρόπο είναι κάτι εξαιρετικά περίπλοκο για του ανθρώπου επιτόπου. Αυτή λοιπόν είναι μια πτυχή που θα πρέπει να εξετάσουμε οπωσδήποτε στην επόμενη μεταρρύθμιση. Δεν πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το μεταρρυθμίσουμε σήμερα, αλλά σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να συμπεριληφθεί στην ατζέντα τη επόμενη μεταρρύθμιση. Το τρίτο ζήτημα που αφορά την απλούστευση, τα προγράμματα, τα προγράμματα αγροτική ανάπτυξη αν τα δείτε και τα συγκρίνετε με τα άλλα προγράμματα, τα προγράμματα αγροτική ανάπτυξης, όπως αν τα συγκρίνετε με τα άλλα ευρωπαϊκά ταμεία Περιφερειακή ανάπτυξης, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα δείτε αμέσως τη διαφορά. Είναι πολύ ογκώδη, πολύ πιο ογκώδη, έχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, ε, ε λεπτομέρειες τόσες που μερικέ φορές φαίνονται υπερβολικέ. Τι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε λοιπόν, να σκεφτούμε λίγο περισσότερο ποιος προγραμματίζει τη στρατηγική. Διότι το τελικό πρόβλημα όταν έχουμε ολοκληρώσει τη σύνταξη των προγραμμάτων είναι ο λεπτομερής κατάλογος των παρεμβάσεων. Οπότε πρέπει να επεξεργαστούμε λίγο παραπάνω τον προγραμματισμό. Και το τελευταίο ζήτημα, για να κλείσω, η ερώτηση που έκανε ο κύριος Ντεκάστρο για, το... για ποιο λόγο δεν έχουμε εθνικά μέτρα. Δεν θα ήταν καλύτερο να είχαμε εθνικά μέτρα. Στην πραγματικότητα αυτό προβλέπεται στον κανονισμό. Τη δυνατότητα να έχουμε ε, μια ομοιομορφία σε εθνικό επίπεδο για τα προγράμματα, ε, για τα κράτη που έχουν πολλά περιφερειακά προγράμματα. Αλλά αυτή η δυνατότητα έχει αξιοποιηθεί ελάχιστα διότι η αξιοποίησή της εξαρτάται από τις σχέσεις εξουσίας που υπάρχουν μεταξύ κράτους και περιφερειών στις διάφορες χώρες. Ε, το να θεσπίσουμε κοινού εθνικούς κανόνες ε, δεν είναι κάτι που είναι σε όλες τις περιπτώσεις αποδεκτό από όλες τις περιφέρειες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουν και οι περιφέρειες κάποιο περιθώριο, κάποια ανεξαρτησία γιατί κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητε. οπότε πρέπει να υπάρχει κάποιο περιθώριο αυτονομίας, ανεξαρτησία για τα επιμέρους περιφερειακά προγράμματα. Ευχαριστούμε. Μπορείτε να απαντήσετε τώρα εν συντομία στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Τρία κυρίως θέματα για να απαντήσω στις ερωτήσεις των Κροατών και των εκπροσώπων του Ηνωμένου Βασιλείου κατανοώ την κατάσταση στην Κροατία, διότι βοήθησε και την Μαλτέζικη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων. Τα προβλήματα θα είναι σημαντικά και μεγάλο βάρος για τις εθνικές αρχές. Εμάς μας βοήθησε πολύ ο αρμόδιος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργάστηκε μαζί μας για να βρούμε λύσεις. Αυτός ο τρόπος λοιπόν είναι σημαντικός. Σε ό,τι αφορά την ονοματολογία των προγραμμάτων ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι αληθές ότι δεν είναι αυτονόητο τι σημαίνουν τα διάφορα μέτρα. Αυτά τα μέτρα που αναφέρατε είναι τα παλιά περιβαλλοντικά μέτρα τα οποία χρηματοδοτούμε ήδη από τη δεκαετία του 1980, δηλαδή για να μπορούν να κάνουν οι αγρότες κάτι που να ωφελεί το περιβάλλον. Και η ανθεκτικότητα της ε, γεωργικής εκμετάλλευσης έχει σχέση με το οικολογικό κίνημα στην Γαλλία. Χρήση δηλαδή νέων τεχνολογιών και νέων τεχνικών για την καλλιέργεια του εδάφους και να κατανοήσουμε τις διασυνδέσεις μεταξύ της καλλιέργειας του εδάφους και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος που παράγεται και από το ίδιο το έδαφος. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στον τομέα αυτό και θα υποφεληθούν πολύ οι αγρότες και οικονομικά και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ενισχυών για το περιβάλλον. Η ε, ενίσχυση, η υποστήριξη των νέων γεωργών πολλά προγράμματα έχουν διοχετεύσει κονδύλια στην στήριξη νέων αγροτών. Με διαφορετικού τρόπου όμω. Και αυτό νομίζω είναι σωστό γιατί στι διάφορε χώρε μέλη τα εμπόδια για την αντικατάσταση, για την εναλλαγή των γενεών στην γεωργία είναι διαφορετικέ. Και συχνά εξαρτώνται από την ε, ε, εθνική οικονομική πολιτική και το γίνεται γενικότερα στην οικονομία. Συχνά οι νεαροί γεωργοί δεν ασχολούνται με τη γεωργική οικονομία διότι τους προσελκύουν άλλοι τομείς ή <clears throat> διότι υπάρχουν σημαντικές ε, απαιτήσει κεφαλαίου για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ε, ανάληψη γεωρικής εκμετάλλευσης. Μέτρα προβλέπονται πάντω στον κανονισμό για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν. Είμαι λοιπόν σχετικά αισιόδοξη από την άποψη αυτή ότι τα διάφορα προγράμματα επιδιώκουν την επίτευξη του στόχου αυτού. Τελευταίο σχόλιο για την απλούστευση. Εδώ ανησυχώ κάπως για τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσατε στα όσα είπα για την απλούστευση. Η απλούστευση δεν σημαίνει μείωση του αριθμού των μέτρων ή μείωση των επιλογών που είναι στη διάθεση των χωρών μελών για τα όσα θέλουν να πράξουν στο τοπικό επίπεδο. Η Ευρώπη έχει τεράστια ποικιλία. Οι δε προκλήσει στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικέ ανά τόπο και ανά χώρα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια εύκαμπτη εργαλειοθήκη που να μπορεί δηλαδή να επιτρέπει την χρήση από διάφορες χώρες διαφορετικών εργαλείων. Αρκεί να υπάρχει ένα κοινό σύνολο προτεραιοτήτων. Εάν μειώσετε στο μισό τα μέτρα, στην ουσία δεν είναι τα χέρια των ανθρώπων που ε, δεν μπορούν να κάνουν πια αυτά που χρειάζεται. Αυτό που με ανησυχεί εμένα στην περιπλοκότητα είναι περισσότερο η περιπλοκότητα των γραφειοκρατικών, των διοικητικών διαδικασιών, των ελέγχων, της υποβολής ε, εκθέσεων και αναφορών και ούτω και αυτό βαρύνει και τις ε, εθνικές διοικήσεις. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ένας κανονισμός μόνο 6 μέτρα θα διευκολυνεί γιατί δεν θα αντικατοπτρίζει όλες τις ανάγκες των χωρών μελών. Χρειάζονται ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στο τοπικό επίπεδο. Να μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή επιτόπου να πει «Κοιτάξτε, έχω μια εργαλειοθήκη, παίρνω λοιπόν το σωστό εργαλείο για να αντιμετωπίσω τη σωστή κατάσταση, την συγκεκριμένη κατάσταση» και όχι να χρειάζεται να συμπληρώσω σελίδες επί σελίδων για να αιτιολογήσω την επιλογή που κάνω ώστε να πείσω κάποιον από το κέντρο ότι είναι ο σωστός τρόπος. Αυτή είναι η απογοήτευση που αισθάνονται πολλές διαχειριστικές αρχές, ότι εν τέλει ανησυχούν διότι δεν μπορούν να δαπανίσουν τα κονδύλια. Και λένε λοιπόν, ε, τότε δεν θα κάνουμε τα περιπλοκά, θα κάνουμε ό,τι είναι πιο απλό. Αλλά δεν είναι αυτό το νόημα του κανονισμού. Όταν μιλώ λοιπόν για απλούστευση, δεν εννοώ μείωση του πεδίου εφαρμογή του κανονισμού, ενώ απελευθερώστε τον μηχανισμό, κάντε τον πιο εύχριστο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σχόλιο του συναδέλφου μου εδώ εξ αριστερών για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα περιφερειακά ταμεία. Δεν χρειάζονται τόσο detailed reporting, τόσο λεπτομερείς υποβολές αναφορών. Πρέπει να βελτιωθεί το πλαίσιο για να εργαστούν και να συνεργαστούν στο τοπικό επίπεδο. Χρειάζεται βέβαια να κινηθούν και οι δύο πλευρέ για να είναι εξασφαλισμένη η σωστή χρήση των κονδυλίων και να μην υπάρξει κατάχρηση χωρίς να αποθαρρύνουν οι άνθρωποι από το να εκμεταλλευτούν το δυναμικό που τους δίνεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις εξηγήσεις που μας δώσατε και όπως είπατε όλα αυτά τα στοιχεία βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Και εμείς ε, ε, που γνωρίσαμε την πρώτη γενιά των ηγετών, όπως ε, σωστά είπατε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επιφέρουμε απλούστευση στα διάφορα δυναμικά στάδια της εφαρμογής και να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Γιατί είδαμε και θετικά στοιχεία και σημαντικούς μοχλούς, αλλά και αρνητικά και υπερβολική επικάλυψη των ελέγχων, η συσσόρευση των ελέγχων. Κάτι που αποβαίνει βάρο ε, της ανάπτυξη ε, της υπαίθρου. Ευχαριστώ πάντως και για τη μελέτη και για την παρουσίαση και για τι απαντήσει που μα δώσατε. Ολοκληρώνεται η δημόσια συνεδρίαση. Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε όσοι δεν δικαιούνται να παραβρίσκονται, παρακαλώ να αποχωρήσουν. Η συνέχεια στις 3 με την δημόσια κρόση για τη ζάχαρη. Ο κύριος Φλάναγκαν. Μπορώ να θέσω μια ακόμη ερώτηση. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Αλλά με μπέρδεψε κάτι που είπατε. Μπορώ να υποβάλω μια ακόμη ερώτηση ή τελειώσαμε δεν μπορείτε να την υποβάλλετε διμερώς αργότερα, γιατί έχουμε πρόβλημα με τη διερμηνία. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δεν μπορείτε, δεν μπορείτε να θέσετε την ερώτηση. Καλώς, αυτό θα κάνω. Σας ευχαριστούμε. Ακολουθεί συνεδρία